Schönen guten Morgen. Καλημέρα. Μπορούμε να αρχίσουμε νομίζω. Οι αποφάσεις των συντονιστών από χτες ε, έχουν ήδη μοιραστεί και αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση μέχρι τις 12.30 εγκρίνονται. Περνάμε τώρα στον τεχνικό πυλώνα του τέταρτου σιδηροδρομικού πακέτου, σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση και ξεκινάμε με την διαλειτουργικότητα. Να κάνουμε έναν έλεγχο πρώτα. Άρχεται η ψηφοφορία. Die Abstimmung ist Geschlossen. Πέρασε. Ωραία. Όλα εντάξει λοιπόν. Wir kommen dann zur Abstimmung über Interoperabilität. Ψηφίζουμε την Κύριε Πρόεδρε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με καλή την πίστη και μέσα σε κλίμα συνένεσης. Θα ήθελα από σήμερα, παρά το γεγονός ότι χθες οι συντονιστές δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε μια απόφαση που να βελτιώσει την κατάσταση εδώ, αλλά τι να κάνουμε έτσι έχει η ζωή για να μπορέσουμε λοιπόν να υποστηρίξουμε κάποια λύση μετά από αυτά τα οποία ανέφερε και η κυρία Μπιλμπάου για να βελτιώσουμε και τη σχέση μας με το Συμβούλιο και με την ελπίδα ότι η Επίτροπος κυρία Μπούλτς θα τηρήσει την υποσχέση που μας είχε δώσει να έρθει ενώπιον του Κοινοβουλίου με ένα πακέτο για την ασφάλεια και για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στον σιδηροδρομικό τομέα. Εγώ θα αποσύρω τις τροπολογίες μου σήμερα το πρωί με την ελπίδα όμως ότι το Συμβούλιο θα διατηρήσει ενωμένο το πακέτο και επίσης ότι θα υπάρξει συνένεση μεταξύ των συναδέλφων. Αλλιώ δεν θα κάνουμε καμία καλή, δεν θα δώσουμε καμία υπηρεσία στο συνδρομικό τομέα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αποσύρω τι τροπολογίε μου. Ευχαριστώ. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Ονομαστική. Ψηφίστε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 38 υπέρ 3 κατά 2 αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Μπιλμπάου. Το επόμενο. Ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Αρχίεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τριάντα υπέρ ε, τέσσερις κατά δύο εποχές εγκρίνεται. Και εδώ ευχαριστώ τον εισηγητή. Ελεύθερος είστε. Λοιπόν, Ευρωπαϊκός οργανισμός της Ρευρωμονάρχης της 38 υπέρ 2 κατά 2 αποχές. Εγκρίνεται επίσης. Περνάμε άρα στην επόμενη ψηφοφορία, συμφωνία με το Μακάο. Δεν είναι ονομαστική αυτή η ψηφοφορία. Και αυτή. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν.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 Κάνουμε εδώ πέρα έλεγχο των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων όσον αφορά το μέσο συνδέοντα στην Ευρώπη. Τα μέτρα αυτά αφορούν το πρόγραμμα εργασίας 2016 για την εφαρμογή του προγράμματος συνδέοντας στην Ευρώπη και τις ε, συνέργειες μεταφορών ενέργειας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 το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το μέσο συνδέοντα στην Ευρώπη. Die Aufrufe zur Einreichung von Vorhaben, die Synergien zwischen den Bereichen Verkehr und Energie erzielen, sowie um die Fortschreibung des Mehr Οι συνέργειες μεταφορών και ενέργειας και το αναθεωρημένο Polites πρόγραμμα για την οικονομική στήριξη να τελειώσει εδώ πέρα πως για μας η εξέταση των προτάσεων της Κομισιόν είναι πάρα πολύ σημαντική. Ειδικά ο κανονισμός αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικό νομοθέτημα για την Επιτροπή μας. Είναι η υποχρέωσή μας να ελέγξουμε πώς εξασκεί η Κομισιόν τις αρμοδιότητες που τους έχουμε παραχωρήσει ως νομοθέτους. Το Tran Committology Newsletter υπάρχει μόνο 8 και 9 μας έχει ενημερώσει για τις αποφάσεις και χαίρομαι που ήρθε εδώ πέρα η Κομισιόν για να μας ενημερώσει για το πώς έχουν τα πράγματα. Ο κύριος Ολιβιέ Ονιδί λοιπόν έχει τον λόγο. Ευχαριστώ. Thank you, Chair, for, for this introduction. Σας ευχαριστώ για αυτή την ε, παρουσίαση. Ευχαριστώ για τις ε, σαφείς ψηφοφορίες που είχατε για το τέταρτο συνδεδομικό πακέτο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στα θέματα αυτά. Για το Connecting Europe Facility θα θυμόσαστε ότι το 2015 είχαμε δεσμεύσει ένα σημαντικό ποσό σχεδόν 13 δισεκατομμύρια ευρώ για 263 συμφωνίες χορήγησης. Ποια είναι τώρα η κατάσταση σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό για να μπορέσουμε να το δούμε στα πλαίσια των ε, τροποποιήσεων στο πρόγραμμα εργασίας που έχετε ενώπιόν σα. Έχουμε κλείσει τη δεύτερη πρόσκληση βάσει του Connecting Europe Facility. Στις 16 Φεβρουαρίου έκλεισε αυτή η πρόσκληση και είναι σαφές ότι είναι πολύ περισσότερες αιτήσεις από τη δυνατότητα χρηματοδότησης 7,6 δισεκατομμύρια ευρώ προβλεπόταν για αυτή την πρόσκληση, 1,1 για, τον γενικό, ε, για το γενικό πλαίσιο και 5,6 μέσα στα πλαίσια το, των κονδυλίων συνοχής. Πιστεύουμε ότι όλες οι απαραίτητες, όλες οι διαθέσιμες μαλοχρηματοδοτήσεις θα χρησιμοποιηθούν. Αυτό δεν μας αφήνει πολύ περιθώριο ελιγμών τα επόμενα χρόνια, εκτός φυσικά αν προχωρήσουμε σε κάποιες ενεργητικές αποφάσεις, κάτι το οποίο θα σας παρουσιάσουμε ως ονουπό. Η κατάσταση λοιπόν για τα προγράμματα εργασίας που έχετε ενώπιόν σας, έχετε τέσσερα τέτοια προγράμματα. Ένα είναι το ετήσιο πρόγραμμα διαφορετικού ε- είδους, <clears throat> είναι ένα πρώτο πείραμα μέσω του οποίου είναι δυνατόν με τη νέα νομική βάση της, ε, του Connecting Europe Facility να εφαρμοστεί. Ήταν κάτι που ζήτησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ουσιαστικά για να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε σχέδια που έχουν χαρακτήρα συνέργειας μεταξύ των μεταφορών και της ενέργειας. Αυτό είναι το πρώτο λοιπόν πρόγραμμα εργασίας. Το δεύτερο αποτελεί ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για τις μεταφορές. Το τρίτο είναι το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για τα ε, μέσα δανειοδότησης για το Connecting Euro Facility και επίσης υπάρχει το πρόγραμμα εργασίας για το πολιετές ε, σχέδιο για την υποστήριξη δραστηριοτήτων. Όλα αυτά με πιο απτό τρόπο θα οδηγήσουν σε δύο πρόσθετες προσκλήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος για προτάσεις που θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο του 2016. Καταρχήν η λεγόμενη πρόσκληση για συνέργειες μεταξύ μεταφορών και ενέργειας για συνολικό ποσό 40 εκατομμυρίων, μια δεύτερη πρόσκληση για τις μεταφορές για 90 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια στο πλαίσιο της συνοχής για τα σχέδια μέσα στο κεντρικό δίκτυο που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1 και 40 εκατομμύρια μέσα στο γενικό πλαίσιο χρηματοδότησης για δύο προτεραιότητες οι οποίες δεν συμπεριλήθηκαν στην προηγούμενη πρόσκληση που μόλις έκλεισε, οι εμπορευματικές υπηρεσίες και τα θέματα του θορύβου στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Η τρίτη τροποποίηση του προγράμματος εργασίας θα μας επιτρέψει να υποστηρίξουμε για 66 εκατομμύρια ευρώ ε, να υποστηρίξουμε τα καινοτόμα ε, εργαλεία βάσει του μέσου δανειοδότησης του ΣΕΦ και το τέταρτο που είναι πολυετές καλύπτει 80 εκατομμύρια και προβλέπεται να χρηματοδοτήσει δράσεις υποστήριξης σε δραστηριότητες όπως είναι το ΣΕΖΑΡ, το EITS, οι διάδρομοι για τις εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές και τα θέματα πλοήγησης. Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον. Συνολικά, θα έχουμε πια στο μέλλον ένα περιορισμένο μονάχα ποσό κονδυλίων, 3 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος της ε, περίοδου πολιετούς ε, δημοσιονομικής ε, σχεδίασης. 1,6 δισεκατομμύρια επί τη βάση χορηγήσεων που όμως έχουν προσδιοριστεί για τα τελευταία χρόνια της, των τωρινών δημοσιονομικών προοπτικών και επίσης 1,6 περίπου δισεκατομμύρια τα οποία καταρχήν προβλεπόσταν για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για το Connecting Europe Facility. Ως εκ τούτου εξετάσουμε τους διάφορους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε την υποστήριξη σχεδίων και στο άμεσο μέλλον. Είδαμε ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον όπως φάνηκε στη δεύτερη πρόσκληση ενδιαφέροντος που είχε πάρα πολλές αιτήσει και βλέπουμε να υπάρχει θετική πρόοδος για το σύνολο των διευρωπαϊκών το σχεδίο για τα διευρωπαϊκά δίκτυα που είναι κάτι το οποίο σας έχουν αναφέρει κατ' επανάληψη συντονιστές των TNT. Και ποιες είναι τώρα οι προ... προοπτικές για το μέλλον και οι επιλογές μας. Εμείς από του χρόνου θα είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε κάποια από τα κονδύλια τα οποία δεν είχαν εκταμιευτεί από αυτούς οι οποίοι έχουν παρουσιάσει σχέδια. Θα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τη διαδικασία use it or lose it. Τα, οι πρώτες δόσεις θα καταβληθούν του χρόνου. Δεύτερον, πιστεύουμε ότι κατά ψευτανότητα υπάρχει σημαντικός αποχρόν λόγος για να μπορέσουμε να προτείνουμε μία μεταφορά από τα χρήματα τα οποία προβλεπόταν για τα χρηματοδοτικά εργαλεία προς την γενική γραμμή του προϋπολογισμού, κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να δώσουμε χορηγήσεις προς σχέδια. Έχουμε τώρα το, τη διευκόλυνση EFSI, e δηλαδή το Ταμείο Juncker, και θα υπάρξει μια κανιβαλικού χαρακτήρα σχέση μεταξύ των δύο διευκολύνσεων. Και στα πλαίσια της ε, αναθεώρησης των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών θα προσπαθήσουμε να εμπροστοφορτήσουμε τις ε, ε, ε, τρέχουσες ανάγκες χρησιμοποιώντας κονδύλια τα οποία προβλεπόταν για το τέλος της ε, δημοσιονομικής περίοδου ώστε να έχουμε την δυνατότητα ήδη από του χρόνου να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις προτεραιότητε. Εν τέλει, δεδομένης της μαζικής επιτυχίας της ε, μεταφοράς του λεγόμενου συνολικού ποσού για την συνοχή που μεταφέρθηκε στο Connecting Europe Facility, Μία από τις επιλογές μας θα μπορούσε να είναι να δούμε αν μέσα στα πλαίσια των διαφορετικών ταμείων θα υπήρχε λόγος εισαγωγής και πάλι μέσα στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεώρησης των πολιετών προοπτικών να κάνουμε και πάλι μια περαιτέρω μεταφορά χρηματοδοτικών μέσων προς το CEF, το Connecting Europe Facility. Αυτό φυσικά θα είχε μεγάλη επίπτωση γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ήδη από του χρόνου μια νέα πρόσκληση. Πιστεύουμε ότι μια τέτοια πρόσκληση θα είχε μεγάλη σημασία, μεγάλο ενδιαφέρον με τρεις προτεραιότητες που έχουμε προς το παρόν στο μυαλό μας. Η πρώτη θα ήταν να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα συνολικό ποσό το οποίο μπορεί να δοθεί υπό μορφή χρήμα χορηγήσεων αλλά για τις ε, μικτές λεγόμενες ενέργειες, δηλαδή υποστήριξη σχεδίων που θα είναι συγχρόνως επιλέξιμα επί τη βάση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως είναι το EFSI ή άλλων σχεδίων, ώστε να γίνουν όλα αυτά τα σχέδια πιο ελκυστικά στους ιδιωτικούς επενδυτές, ιδίως σε δύσκολες περιοχές όπως το ΣΕΖΑΡ, παραδείγματος χάρη, ή η εσωτερική υδάτινη δρόμη. Μια περαιτέρω δυνατότητα θα είναι, όπως ξέρετε κύριε Πρόεδρε, έχουμε αναλάβει δράση στο να εξετάσουμε τους μικρούς ελείποντες κρίκους από το συνολικό δίκτυο. Στην Επιτροπή σας εσείς έχετε τονίσει κατ' επανάληψη ότι πέραν των μεγάλων σχεδίων θα έπρεπε να εστιάσουμε και σε μερικά μικρότερα τμήματα, μικρούς κρίκους οι οποίοι ελείπουν από το πλήρες δίκτυο, ώστε και εκεί να μπορέσει να υπάρξει μια σημαντική βελτίωση και δημιουργία νέας ικανότητας. Ε, κυρίως φυσικά στις ιδοδομικές δράσεις. Η δεύτερη λοιπόν προτεραιότητα για μια πρόσκληση θα μπορούσε να είναι ακριβώς να στοχοποιήσουμε καλύτερα από τους ελείποντες κρίκους επί τη βάση του αναλυτικού έργου που έχουμε φέρει σε πέρας μέχρι τώρα και που ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε ταχαίως να σας παρουσιάσουμε και τρίτη προτεραιότητα θα είναι η καινοτομία. Γιατί εδώ η καινοτομία πρέπει να αντιμετωπιστεί ευρία τη ενία. Βλέπουμε πολλές δυνατότητες να χρησιμοποιηθεί η καινοτομία στα εναλλακτικά καύσιμα, στα νέα συστήματα διαχείρισης ροών, στο συνδρομικό τομέα, αλλά επίσης και στην επίτευξη λύσεων στους αστικούς χώρους. Αυτό το τμήμα λοιπόν θα έπρεπε και αυτό να τύχει περαιτέρω ενίσχυσης στη χρηματοδότησή του μέσα στα πλαίσια μιας νέας πρόσκλησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος για την παρουσία σας και για τα λεγόμενά σας. Θα δώσω τώρα το λόγο πάλι στους συντονιστές πρώτα απ' όλα στον Μάρκους Πίπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για την τοποθέτηση αυτή, για την πρόοδο του ΣΕΦ. Πραγματικά θετικά αυτά τα οποία μας είπε και δεν μας προξενεί η έκπληξη. Εμείς θεωρούμε ότι το μέσο ενδιαφέροντας στην Ευρώπη είναι πολύ θετικό και καταφέρνει να βρει έργα να τα συνδέσει με χρηματοδότηση όταν έχουμε επίσης νέες ιδέες όπως τώρα όπου μπορούν τα σημαντικότερα πράγματα να γίνουν με λίγα λεφτά είναι κάτι το οποίο χαιρετίζουμε. Όμως παραμένει ένα ερώτημα προς την Κομισιόν το οποίο αφορά τον προϋπολογισμό του 2016. Έχουμε ένα ζήτημα αρχής για το τι κάνει η Κομισιόν εδώ πέρα. Έχουμε υποσχεθεί πως όταν υπάρχουν περιθώρια στον ετήσιο προπολογισμό τα λεφτά το ΣΕΦ θα τα λαμβάνει πίσω για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει και τις εγγύησεις ε, του ΕΦΣΙ. Είναι δικά μας τα χρήματα και μας είχαν υποσχεθεί ότι θα ε, επιστρέφονται όταν είναι αδιάστα. Τώρα όμως κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του 2016 είναι το εξή. Η Κομισιόν ήρθε με μια διαπραγματευτική θέση που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ευτυχώς είναι αυτά τα 150 εκατομμύρια τα οποία είναι πάλι διαθέσιμα για το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη και τον ορίζοντα 2020 αλλά πέρα από αυτό το ορίζοντας 2020 έχει άλλα 40 εκατομμύρια τουλάχιστον 40 εκατομμύρια και άλλα επιπλέον για το εράσμος και το κόσμο και το ερώτημα προς τους εκπροσώπους της Κομισιόν είναι αν είναι απαραίτητο αυτό για το μέσο συνδέοντα στην Ευρώπη μας είπαν όχι έχουμε αρκετά λεφτά για τα έργα τα οποία έχουν υποβληθεί. Έτσι μας το είπαν καταλήξει και τώρα δεν καταλαβαίνω πώς με μια τέτοια θέση μπορεί κάποιος να πάει σε οικονομικές διαπραγματεύσεις, γιατί ξέρουμε πως ο πρώτος διαγωνισμός, τα 12 δισεκατομμύρια, έχει αιτήσει ε, για 37 δισεκατομμύρια. Το τριπλάσιο δηλαδή. Πώς μπορεί η Κομισιόν λοιπόν να μας λέει ότι δεν χρειάζονται επιπλέον χρήματα. Αυτό μας απογοήτευσε. παίρνει από τέσσερις μήνες είχα γράψει μία επιστολή στην κυρία Μπούλτς, καμία απάντηση δεν έλαβα. Μετά προσπάθησα μέσω του συντονιστή, του Βίμ Φαντεκάμπ και κάποιον άλλο από τη γερμανική ομάδα. Ξανά γράψαμε την ίδια επιστολή προς την κυρία Επίτροπο, πάλι καμία απάντηση. Ε, και τώρα προσπαθούμε να εμπλέξουμε την Επιτροπή και ελπίζουμε να δούμε το πώς ε, διαπραγματεύεται η Κομισιόν και να δούμε και τη διαπραγματευτική ομάδα να ρίξει λίγο φως ε, στην υπόθεση γιατί δεν γίνεται να υπάρχει τόσο μεγάλη προτίμηση στην πλευρά της έρευνας και β όταν ρωτάμε την Κομισιόν να μας λέει πως ε, είναι όλα εντάξει και έχουν κρίνει όλα τα έργα ικανοποιητικά. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει εδώ πέρα ξεκάθαρα η Κομισιόν τι γίνεται. Και πώς βλέπει και τα επόμενα έτη για τις πολιετήσεις δημοσιονομικές προοπτικές. Θα τα δεχτούν παθητικά ή θα φροντίσει η Κομισιό, θα φροντισει η κομισιον κάποτε. Σας ευχαριστώ. Τα συζητήσαμε αυτά χτες ε, και στην ε, συνεδρίαση των συντονιστών και οπωσδήποτε θα δώσω συνέχεια εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής. Ντομινίκ Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ την Κομισιόν για την ε, εξήγησή της. Θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, για τις πιστώσεις του Connecting Europe Facility. Η ανακύκλωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί νέο χρήμα. Απλώς απελευθέρωση χρημάτων μετά από δύο χρόνια. Η αναπροσαρμογή ή η ανακύκλωση είναι ουσιαστικά κινητοποίηση κονδυλίων από τα διαφορετικά ταμεία προς το CEF. Εμείς δίνουμε μάχη για να πετύχουμε μια πραγματική αναθεώρηση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου, τόσο ώστε να δοθούν πραγματικά χρήματα στο ΣΥΕΦ. Γιατί έχει μια τεράστια επιτυχία. Δεν το υπενθυμίσατε, αλλά θα μπορούσατε να είχατε πει πόσε ήταν οι προτάσει σε σχέση με τον αριθμό των ε, έργων που επιλέχθηκαν τελικά. Συνήθω είναι διπλάσιε ή τριπλάσιε οι προτάσει. Ε, υπάρχουν δηλαδή πληθώρα προτάσεων που δεν χρηματοδοτούνται τελικά, που δεν επιλέγονται. Ε, το ότι δεν χρηματοδοτούνται σημαίνει ότι δεν υλοποιούνται. Γιατί υπάρχουν πολλές δυσκολίες να κινητοποιήσουμε στον τομέα των μεταφορών κονδύλια. Μέχρι στιγμής οι μηχανισμοί επενδύσεων τύπου ΕΦΣΙ του σχεδίου Juncker για λόγους που έχουν να κάνουν με τη φύση των έργων και την απουσία κερδών ε, επί των επενδύσεων ε, δείχνει ότι δεν μπορούμε να προωθήσουμε αυτά τα έργα. Στην πραγματικότητα πρέπει να κόψουμε τους δύο μηχανισμούς, να τους αποκόψουμε μεταξύ τους. Η Κομισιόν θα πρέπει να πει ξεκάθαρα, ίσως φέτος το 16 ή το 17, ποιο είναι το ποσοστό των ε, ταμείων του Connecting Europe Facilities που χρηματοδοτούνται είτε με ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε μέσω του ΕΦΣΥ του σχεδίου Juncker δηλαδή. Τι είδους ε, χρήματα πήρατε από το ΕΦΣΥ επιπροσθέτως πέρα από αυτά που δίνει το CEF. Είναι πολύ σημαντικό το ξέρουμε αυτό γιατί θα πρέπει να φτάσουμε σε μια οικονομική πρόβλεψη προκειμένου να φτιάξουμε ένα νέο μηχανισμό ή να αναπροσαρμόσουμε αυτό το μηχανισμό. Πόσα χρήματα πήραμε από το ΕΦΣΕ για να πάνε στο ΣΥΕΦ, θέλουμε να το ξέρουμε αυτό. Επίσης, βλέπουμε ότι επειδή δεν έχουμε πολλά χρήματα για τις οριζόντιες προτεραιότητες, τελικά πάσχουμε ε, στην πραγματικότητα ε, για, τις, για την ενέργεια, για τα δίκτυα, για την ψηφιακή αγορά και για την, ε, το δυναμικό εναλλακτικής ε, το δυναμικό ανάπτυξη αναλυτική ενέργεια που είναι προτεραιότητε τη Κομισιόν, δεν μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά. <clears throat> Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν κάποιε σωστέ προβλέψει σε οικονομικό επίπεδο. Θέλω να θέσω μια ερώτηση προ την Κομισιόν. Εκτιμάτε. ότι μπορούμε να απελευθερωθούμε από τα παρατήματα για να πάμε προς ε, διαφορετικές επιλογές. Παράδειγμα, αν πάμε, πάρουμε τους ελίποντες κρίκους που αναφέρατε, αυτοί οι ελίποντες κρίκοι βρίσκονται στο... θα πρέπει να τους αναζητήσουμε στο παράρτημα 1 ή εκτός αυτού του παραρτήματος ή εκτός και των άλλων δύο παραρτημάτων. Τέλος, όπως είπε και ο Μάρκους Πίπερ, θέλουμε η Κομισιόν να μιλήσει ξεκάθαρα και στα πλαίσια του ετήσιου προπολογισμού, κυρίω για την ανθεώρηση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου, θέλω να σα πω ότι η θέση του Συμβουλίου δεν είναι και τόσο ενθαρρυντική, καταρχήν τουλάχιστον. Εμεί πιστεύουμε ότι θέλουμε μια πραγματική αναθεώρηση. Την έχουμε ανάγκη. Μην ξεχνάτε και κάποιες εθνικές ε, εκλογές μπορεί να παίξουν κάποιο ρόλο για το πώς θα επηρεάσουν αυτές το δημοσιονομικό πλαίσιο ε, δεν θα πρέπει να περικόπτουμε αυτά τα κονδύλια. Ε, κρίμα, κρίμα που κάποια από αυτά τα κονδύλια ε, πήγανε για άλλους σκοπούς. Ε, κονδύλια που τα είχαμε για το CEF, για το Connecting Europe Facility και για τις δικές μας προτεραιότητες. Ιζαμπέλα Ντεμόντε. Θετικές είναι αυτές οι παρατηρήσεις, γιατί πιστεύω ότι όλα αυτά που ακούστηκαν σε σχέση με τις προτεραιότητες της τρίτης ζώνης είναι προτεραιότητες ε, που μου όλους σύμφωνους. Ιδίως για τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων με το ΕΦΣΥ. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ε, αυξάνουμε το, τις επιπτώσεις του Connecting Europe Facility και εξασφαλίζουμε την ε, ανάπτυξη. Ε, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τους ελείποντες ε, κρίκους. Ε, ας πούμε, η Ιταλία, Σλοβενία. έχουμε δύο διαφορετικές ιδεοδομικές γραμμές, οι οποίες δεν, χρησιμο, δεν συνδέονται καθόλου. Δεν υπάρχει σημείο τομή, α πούμε, και επομένω είναι χρησιμοποιείται. Δηλαδή, ουσιαστικά πάνε στράφη, α πούμε θα πρέπει project τα οποία ξεκίνησαν στο παρελθόν και αυτά που θα αρχίσουν στο μέλλον μέσω αυτών των ε, έργων ε, να προχωρήσουν. Επίσης, ε, θα πρέπει να συνδέσουμε και τα διάφορα εσωτερικά λιμάνια. Υπάρχουν εκεί τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Και το ερώτημα μου είναι, λαμβάνετε υπόψη και, την, και τον τουρισμό ε, όταν αξιολογείτε αυτές τις, αυτούς τους διαγωνισμούς, αυτές τις προσφορές. Γιατί πάντα όταν μιλάμε ας πούμε για, μια, για, για κάποια έργα λέμε «Α, ας πούμε το τάδε λιμάνι έχει τέτοια δυνατότητα μεταφοράς ε, φορτίου ας πούμε». Αλλά δεν είναι μόνο το φορτίο, είναι και ο τουρισμός. Πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Κυρία Ντέλη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Νίδη για την παρουσίασή σας. Έχω πολλαπλές ερωτήσεις. Θέλω να επανέλθουμε καταρχάς σε αυτό το μεγάλο αχρίαστο έργο το Νοτούρα. Ποιες θα είναι οι δημοσιονομικές γραμμές που θα δοθούν εκεί γιατί έχει τεράστιες χρηματοδοτικές ανάγκες αυτό το έργο. Αυτή τη βδομάδα έγινε μια γαλλο-ιταλική σύνοδος κορυφή που ήταν το εναρτήριο λάκτισμα ουσιαστικά για τις, α, ε, τους διαγωνισμούς των σχετικών έργων. Ακούστηκε ότι το κόστος όμως θα είναι 8,4 εκατομμύρια ευρώ και θα έχει σαν στόχο να ξεκινήσουν οι εργασίες για αυτό το έργο αυτό αλλά μας λένε ότι λόγω της επέκτασης των ε, κονδυλίων είναι 40% αυτά που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας, μας λένε ότι θα φτάσουμε τελικά στα 10 εκατομμύρια λόγω του κόστους των πρώτων υλών και του πληθωρισμού κτλ. κτλ. Κομισιόν, ερώτημα η, τα κέρδη για τέτοιου τύπου επενδύσεις ε, είναι ικανοποιητικά σε ό,τι αφορά τη, ε, τη δημιουργία θέσεων ε, απασχόλησης, την ε, ε, συμμετοχική δημοκρατία, μια, μια και είναι ένα έργο στο οποίο συμμετέχουν και οι πολίτες κτλ. Επίσης, το θέμα αυτό μπορεί να συνδέεται με το ποιος λαμβάνει αυτή τη βοήθεια. Μας εγγυάστε ότι θα ελέγξετε το ευρωπαϊκό δημόσιο χρήμα και ότι θα πάει στις τσέπες των μαφιόζων. Πού δεν θα χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά τα κονδύλια, φυσικά. Δεύτερον, κύριε Νίντι, είπατε ότι η Κομισιόν εκτιμά ότι αύριο μεθαύριο θα χρειαστεί να μετακινηθούν χρήματα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Γιατί δεν μας δίνετε σήμερα χρήματα για την συντήρηση των ισχύων των δικτύων και κυρίως των τρένων. Το χρειαζόμαστε αυτό. Τα κράτη δεν παίρνουν στα σοβαρά υπόψη τις ανάγκες αυτές και θεωρώ ότι η Κομισιόν μετά από την COP21 θα έπρεπε να φτιάξει ένα μεγάλο ευρωπαϊκό project για την ανακαίνιση των σιδηροδρομικών δικτύων, των ισχυών των σιδηροδρομικών δικτύων. Τρίτον, μίλησα για την COP21 και για τη μείωση επομένω του διοξιδίου του άνθρακα, γιατί εκεί πάει το μυαλό μα, Θα ήθελα να μου πείτε ε, το εξή. Κάτι που ενδιαφέρει εμένα και την ε, ομάδα μου, του ψυχολόγου. Μήπως θα πρέπει τέλος πάντων να μπούμε ουσιαστικά στον 21ο αιώνα με μία μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων. Όλοι το είπαν στην COP21. Η Κομισιόν λέει τα δικά της, αλλά πολύ συγκεκριμένα. Όταν μιλήσατε για μεταφορές και ενέργεια, πέστε μου, πού βρισκόμαστε ε, σε ό,τι αφορά την συγκινητικότητα και σε στην εκκίνηση μιας πραγματικής αστικής κινητικότητας βιώσιμης, βιώσιμης όμως. Μπορείτε να μας εγγυήσετε ότι η συγκινητικότητα η αυριανή, η δεν θα έχει μόνο σαν κέντρο το, ηλεκτρον το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά και το ποδήλατο κτλ. Υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε για αυτή τη νέα κινητικότητα, τη συγκινητικότητα. Και αυτή η βιώσιμη αστική κινητικότητα δεν είναι μόνο το ηλεκτρονικό αυτο, αυτοκίνητο. Ποιες είναι οι καινοτομίες σας, ποιες είναι, ποια είναι τα project που θα προωθήσετε, πώς το βλέπετε γενικά. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κάποια ερωτήματα τα οποία πρέπει να τύχουν απάντησης τα είπε κάπως διπλωματικά ο Ντόμινικ Ρικέ ακολουθώντα τον γαλατικό τρόπο έκφραση. Εγώ θα τα πω και πιο ομά, λέει η κυρία Μάισνερ. Για μένα τίθεται το ερώτημα το εξή. Εγώ βλέπω τώρα να γίνεται κάπως παράδοση να βγαίνουν λεφτά από το Connecting Europe και να πηγαίνουν λεφτά στο EFSI. Εγώ πιστεύω ότι τα χρήματα αυτά μετά πηγαίνουν σε άλλες χρήσεις. Νόμιζα ότι είχε ξεπεραστεί αυτή η διαδικασία. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί κάτι τέτοιο. Για το ΕΦΣΥ έχουμε σχέδια τα οποία φυσικά είναι στον τομέα μεταφορών, αλλά δεν είναι μονάχα στον τομέα των μεταφορών. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι για αυτά τα άλλα προγράμματα εμεί δεν έχουμε καμία δυνατότητα επηρεασμού. Πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν αυτέ τι επενδύσει εν γέννη, αλλά τα χρήματα τα οποία βρίσκονται στο ΣΕΦ, στο Connecting Europe, θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν ενέργειες στον τομέα μεταφορών. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω κατά πόσο θα υπάρξει η τροποποίηση αυτών των ενεργειών προς την κατεύθυνση που θέλουμε εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών. Επίσης, τι θα γίνει με τα χρήματα τα οποία δεν θα χρησιμοποιηθούν. Εμείς είπαμε ότι ό,τι χρήματα δίνονται πρέπει να δοθούν σε σχέδια μόνο τα οποία ανταποκρίνονται στις προτεραιότητές μας. Τα χρήματα τα οποία θα περισσέψουν πότε θα επιστρέψουν ή θα χρησιμοποιηθούν κάπου όλο. Φαντερκάμπ. Ευχαριστώ λέω ο κύριος Φαντερκάμπ. Κύριε Πρόεδρε, η θα χρησιμοποιηθουν καπου ολο Κάμπ. ευχαριστω λεω ο κυριος Κάμπ. κυριε προεδρε πρωτη μου ερώτηση ετέθη από την κύρια Γκεζίνε Μάισνερ που λέει πως η αρχή αυτή use it or lose it είναι σημαντική αλλά τι σημαίνει αυτό πρακτικά όπως είπε και η Γκεζίνε μπορείτε να μας πείτε λίγο κάποια πράγματα για πόσα τι επιστρέφεται τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για άλλα έργα δεύτερη ερώτηση για τις πρώτες εμπειρίες με το έύση. Θα έχουμε και άλλους τρόπους μεταφορών όπως την εσωτερική πλοία και τον σιδηρόδρομο γιατί φοβούνται όλοι πως ε, το ΕΦΣΙ θα πάει μόνο στους αυτοκινητόδρομους και όχι για σιδηρόδρομους και εσωτερική πλοία. Υπάρχει τρόπος ε, να συμπεριληφθούν και οι άλλοι δύο τρόποι μεταφορών. Ευχαριστώ. Δεν ακούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια συγκεκριμένη ερώτηση έχω Πόσο έχει προχωρήσει η υλοποίηση των διευρωπαϊκών αξώνων μαζί με το ΣΕΦ και η σύνδεση του ΕΦΣΥ, του σχεδίου Γιούνκερ, για να πάμε σε επενδύσεις στις υποδομές. Καλό θα ήταν η Κομισιόν, ο κύριος Ονίδη, να μας πει πόσο έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Το επόμενο δεν έχουμε μόνο όπως είπαμε τους αυτοκινητοδρόμους της θάλασσας ε, για να μεταβούμε στην ναυτιλία που είναι πολύ σημαντικό να δούμε και την κατανάλωση ενέργειας αλλά υπάρχει και επιβάρυνση του πληθυσμού από τον θόρυβο του σιδηροδρόμου που ειδικά οι εμπορικές αμεξοστοιχίες κάνουν πολύ θόρυβο. Έχουμε κάπου νομίζω διαπραγματευτεί στα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα υπάρχουν πάρα πολλά εθνικά έργα όπως στη Γερμανία ε, να αλλάξει το τροχαίο υλικό ε, πώς λειτουργεί αυτό ο συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ευχαριστώ. Τώρα θα μιλήσω εγώ. Χαίρομαι βεβαίως για το ότι η Κομισιόν κατέληξε στο ότι τα μεθοριακά σημεία πρέπει να έχουν μια προτεραιότητα. Βεβαίω, εντάξει, το ζήτημα δεν είναι μόνο στην Βεσφαλία αλλά και αλλού. Αλλά το θέμα είναι, μπορείτε να δώσετε λεφτά σε συγκεκριμένα έργα. Ξέρουμε πω από το 1990 έχει επιδεινωθεί η κατάσταση στι εκπομπέ γιατί η Κομισιόν έχει επιτύχει μείωση των εκπομπών ε, στην ε, βιομηχανία αλλά ε, συμβαίνει το αντίθετο στις μεταφορές. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις τώρα. Από το Βερολίνο στην Μπρατσλάβα που είναι φέτος η πολιτική πρωτεύουσα της Ευρώπης έστω ότι θέλει να πάει κανείς εκεί πέρα δεν υπάρχουν συνδέσεις βλέπουμε και υποτίθεται ότι τα προωθούμε ότι είναι η πολιτική πρωτεύουσα της Ευρώπης και τι λείπει λείπουν 50 χιλιόμετρα ηλεκτρικού δικτύου, αλλά μονίμως δηλαδή όταν μιλάμε για εξηλεκτρισμό μιλάμε για τα αυτοκίνητα, όχι για το σιδηρόδρομο. Βλέπει λοιπόν η Κομισιόν κάποιες δυνατότητες να πείσει τη γερμανική κυβέρνηση. Περιμένω, ναι. Γιατί ε, δεν ε, κάνετε κάτι τέτοιο, θα σας δώσουμε τα λεφτά. Να ξαναφτιάξετε τη γέφυρα που καταστράφηκε στον πόλεμο. και να τους πούμε ναι για το έργο Erfurt Νιρεμβέργη θα λάβετε ένα δισεκατομμύριο αλλά μόνο εάν υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Το Λιόν Τωρίνο αναφέρθηκε ήδη. Εκεί πέρα ξέρουμε πως αυξάνεται το κόστος και θα απασχολήσει αυτό την Επιτροπή Έλεγχου του Προπολογισμού αλλά μήπως η Κομισιόν έχει τη δυνατότητα να πει ότι ναι θα κρατήσει τουλάχιστον 13 χρόνια. Αλλά αν υπάρξει ανακαίνιση του υφιστάμενου δικτύου, ποιο το κόστος και η διαφορά και η αλλαγή στην ταχύτητα. Για κάντε το αυτό, να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Εγώ θεωρώ πως ε, τα μεγάλα έργα δεν έχουν τόσο μεγάλη σχέση με την... Ε, κίνηση τους ε, δρόμους είναι περισσότερο το λόμπι των εργολάβων. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για αυτό που σας είπα και για να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή. Αυτά τώρα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ για τις ε, ερωτήσεις που δείχνουν νομίζω το ενδιαφέρον που δείχνετε για αυτό το σημαντικό μέσο. Πρώτα στον κύριο Πίπερ, συγγνώμη αλλά δεν έχω δει ούτε την πρώτη ούτε τη δεύτερη επιστολή την οποία αναφέρατε. Οπότε αν μπορείτε να μου τη στείλετε απευθείας θα φροντίσω να λάβετε απάντηση. Πραγματικά δεν έχω δει τέτοια επιστολή. Και θα απαντήσουμε. Ε, για τη γενική χρηματοδότηση. Κοιτάξτε, το ΣΕΦ νομίζω είναι φοβερή επιτυχία, το μέσο συνδέοντας στην Ευρώπη και σαφώς ε, ποτέ δεν θα υπάρχει επαρκής ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οπότε ναι, αν κάποιος συνάδελφός μας ε, σας είχε δώσει κατά λάθο την εντύπωση πως έχουμε επαρκή χρηματοδότηση, προφανώς αυτό δεν ισχύει. Θέμα επεγνωσμένα επιπρόσθετη χρηματοδότηση. και πραγματικά το μέσο αυτό τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και για τις χώρες της συνοχής. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε εκταμιεύσει τόσο γρήγορα τα κονδύλια στο κομμάτι της ε, συνοχής και νομίζω πως οι πρώτες χώρες που θα αποδείξουν την αξία ακριβώς ε, αυτού του μέσου είναι οι χώρες της συνοχής. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε κατά στο πλαίσιο της συζήτησης της ε, μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης. Μετά για την ανακύκλωση, το use it or lose it προφανώς δεν μπορεί να θεωρηθούν ε, σε επιπρόσθετα κονδύλια. Έχει δίκιο ο κύριος Ρικέ. Αλλά τουλάχιστον ο κανόνας αυτός ο οποίος για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί φέτος ελπίζουμε να μας επιτρέψει να ενισχύσουμε, να βελτιώσουμε τον προϋπολογισμό που είναι διαθέσιμος ε, για το επόμενο έτος. Οπότε θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και θα ζητήσουμε από όλους τους αναδόχους να μας πούν πού βρίσκονται οι δαπάνες για να μπορέσουμε να ανακυκλώσουμε ως το δυνατόν περισσότερη χρηματοδότηση για την ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν ε, χρηματοδοτήσεις έτσι ώστε τα έργα των μεταφορών να γίνουν πιο ελκυστικά για ιδιώτες επενδυτές και να υπάρξει μεγαλύτερη ορατότητα στο ΕΦΣΙ είναι ένα πραγματικό ζήτημα. Είναι κάτι το οποίο θα σας προτείνουμε. Βεβαίως, το σκεπτικό δεν είναι τώρα να μπει όλη η διαθέσιμη χρηματοδότηση στο σχέδιο Juncker. Όχι. Σκοπεύουμε να μεγιστοποιήσουμε τη χρήση του σχεδίου στρατηγικών υποδομών για τα έργα μεταφορών, αλλά μια που, αυτά τα έργα είναι ε, υψηλού ρίσκου, νομίζω πως οι επιχορηγήσεις ε, τα κάνουν πιο ελκυστικά. Για την ερώτηση του κυρίου Ρικέ θα σας στείλω ένα κατάλογο παραδειγμάτων όπου έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει επιπρόσθετη χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων για να έχουμε χρηματοδότηση μεγάλης κλίμακας. Ένα από αυτά το ξέρετε πάρα πολύ καλά είναι η χρηματοδότηση του λιμανιού του Καλέ. Οι οριζόντιες προτεραιότητες, αυτό είναι ένα άλλο θέμα νομίζω που αναφέρατε και είναι πράγματι ένας τομέας που δείχνει πόση χρηματοδότηση χρειαζόμαστε για να έχουμε περισσότερες δραστηριότητες στις νέες μορφές κινητικότητας και προσπαθούμε να προωθήσουμε την ε, έγκριση τέτοιων έργων και βεβαίως ε, Μάιο-Ιούνιο θα σας δείξουμε αυτό τα οποία αξιολογούμε αυτή τη στιγμή. Ε, έχουμε πάρα πολύ ελκυστικά έργα στις πόλεις, στα εναλλακτικά καύσιμα, στους νέους τρόπους κινητικότητας που δεν θα μπορέσουμε δυστυχώς να χρηματοδοτήσουμε πλήρως λόγω των γνωστών περιορισμών. Οπότε ε, σαφώς είναι μια προτεραιότητα που θα συνεχίσουμε να τρώθουμε. Όχι μόνο στη φετινή προκήρυξη, αλλά ελπίζουμε να είναι και στην προκήρυξη του επόμενου έτους. Για το παράρτημα τώρα. Το παράρτημα είναι παράρτημα και ο κανονισμός είναι κανονισμός, δεν μπορώ να τα αλλάξω. Αλλά μπορούμε να κάνουμε ό,τι γίνεται μέσω του κανονισμού. Όσον αφορά λοιπόν το περιθώριο αυτό που υπάρχει για να χρησιμοποιήσουμε στο συνολικό δίκτυο έχουμε ακόμα αρκετή ευελιξία. Οπότε θα δώσουμε βάρος ε, στις διασυνοριακές συνδέσεις με βάση την ανάλυση που κάνουμε τώρα, αυτή θα είναι η πρώτη προτεραιότητα και οπωσδήποτε θα ευθυγραμμιστεί με τους περιορισμούς που υπάρχουν όσον αφορά τα ποσά που περιγράψαμε στο παράρτημα. Ε, το ερώτημα της κυρίας Ντελμόντε για τον αντίκτυπο στην ευρύτερη οικονομία ανέφερε τον τουρισμό. Τα περισσότερα έργα που υποβάλλονται σε μας έχουν μια ανάλυση κόστους κόστους-οφέλους και ακριβώς εκεί πέρα δείχνουν το γενικότερο όφελος στην οικονομία, στην τοπική ανάπτυξη και οπωσδήποτε ο τουρισμός είναι μια σημαντική πτυχή. Για το έργο Λιόν Τωρίνο το περίμενα βεβαίως Η χρηματοδότηση είναι γνωστή και είναι επίσης συνέπεια των όσων λέει ο κανονισμός. Για την ώρα έχουμε δεσμεύσει γύρω στα 800 εκατομμύρια. Σας ενδιαφέρει τόσο πολύ, εσάς και άλλους, ώστε σε συγκαιώμαι ότι είναι το έργο το οποίο ελέγχεται περισσότερο από όλα τα έργα τα οποία έχουμε. Κάθε δυνατός έλεγχος ε, ασκείται. Και εμείς το παρακολουθούμε στενά όσον αφορά την υπέρβαση του κόστους που δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής αλλά το παρακολουθούμε οπωσδήποτε για τυχόν αδιάθετα πόσα και τέτοια μεγάλα έργα υποδομών είναι αυτά που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε αυτή την λεγόμενη ανακύκλωση της χρηματοδότησης. Οπότε αυτό το οποίο λέει και η Ανταλή είναι πράγματι θα γίνει και με βάση το Λιόν Τωρίνο για την συντήρηση ε, αποκλείεται ξεκάθαρα από την νομική βάση. Αν θέλετε να αρχίσουμε να χρηματοδοτούμε την συντήρηση, αυτό δεν γίνεται με το μέσο συνδέοντα στην Ευρώπη. Έχουμε κάποια δουλειά που γίνεται με τους ε, συναδέλφους μας. όσον αφορά την ε, ανακαίνιση περισσότερο, όχι την συντήρηση. για ένα τεράστιο σχέδιο ανακαίνησης και η δουλειά που κάνουν νομίζω οι συντονιστές ε, περιλαμβάνει πολλά στοιχεία που θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να αξιολογήσουμε τις ανάγκες και να καταλήξουμε σε κάποιες προτάσεις ε, στο προσεχές μέλλον. Για τα εναλλακτικά κάψιμα ναι, είναι προτεραιότητα. Αν ε, έχουμε περισσότερη χρηματοδότηση θα μπορούσαμε βεβαίω να χρηματοδοτήσουμε περισσότερες λύσεις. Για τα εναλλακτικά καύσιμα. και άλλα μέσα μεταφοράς ε, χαμηλού άνθρακα. Οπωσδήποτε ο Επίτροπος θα σας περιγράψει κάποιες ιδέες που είχαμε για το θέμα αυτό. Οπωσδήποτε θα υπάρχει η πτυχή της χρηματοδότησης και βεβαίως η πτυχή του να γίνουν οι υποδομές μας πιο καθαρές. Και οπωσδήποτε αυτό θα είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε μαζί σας τις ημέρες των διευρωπαϊκών δικτύων. Γιατί είναι ένα από τα θέματα που έχουμε επιλέξει φέτος για το Ρότερνταμ. Για το ΕΦΣΥ. Για να απαντήσω στην κυρία Μάισνα οι μεταφορές απετέλεσαν μια επιτυχία μέσα στο σχέδιο Γιούγκερ στο ΕΦΣΥ. Είναι λάθος να πούμε ότι είμαστε ο πτωχός συγγενής του ΕΦΣΥ, μεταφορές δηλαδή. Τα σχέδια τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί, πάνω από 10 σχέδια μεταφορών στο ΕΦΣΥ, ήδη εκπροσωπούν παραπάνω από το 30% που ήταν το μέγιστο ποσοστό για τον τομέα μεταφορών που είχε προβλεφθεί. Πάμε πολύ καλά λοιπόν στον τομέα των μεταφορών και ελπίζω ότι θα είναι βιώσιμη αυτή η εξέλιξη. Για να είναι βιώσιμη χρειαζόμαστε και περισσότερες χορηγήσεις ώστε κάποια από τα πιο δύσκολα και πιο προτεραιότητα σχέδια να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΦΣΙ. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ΕΦΣΙ. Ξέρετε ότι αυτή η μάχη έχει χαθεί προσπαθήσαμε <clears throat> να εξασφαλίσουμε ότι κάποια από τα κριτήρια επιλεξιμότητας στα διευρωπαϊκά δίκτυα να περιληφθεί στο ΕΦΣΙ. Αυτό δεν έγινε πραγματικότητα στο τέλος, αλλά αυτό το οποίο μπορούμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να συνεργαστούμε με τους συντονιστές, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να υποστηρίξουμε τα σχέδια τα οποία αποτελούν προτεραιότητα για μας και μπορώ να σας πω ότι έχουμε συστηματικά εργαστεί για όλα τα σχέδια που συνδέονται με τους διαδρόμους ώστε να χρηματοδοτούνται συστηματικά αυτά τα προγράμματα από το ΕΦΣΙ. Για τα θέματα θορύβου, κύριε Κούν, στην επόμενη πρόσκληση θα έχουμε 20 εκατομμύρια ακριβώς για τη μείωση του θορύβου στους σιδηροδρόμους. Ελπίζω λοιπόν θα μπορέσουμε να βρούμε και πρόσθετα ποσά τα επόμενα χρόνια, αλλά η λύση δεν μπορεί να έρθει μονάχα με την χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι κάποια από τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει μια θαραλέα προσέγγιση, μια φιλόδοξη προσέγγιση για τη χρηματοδότηση αυτών των σχεδίων. Και στο τέλος του 2015 κάναμε σαφές ότι η προσέγγιση μας θα πρέπει να είναι να επιβάλλουμε την ε, ανασκευή όλων των βαγονιών, των ε, του τροχαίου υλικού με τα σύνθετα αυτά υλικά ώστε να μην ώστε να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι πολύ δύσκολο και πολύ επίπονο σε ορισμένε περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα καταθέσουμε λοιπόν μια πρόταση τεχνικού χαρακτήρα φυσικά, <clears throat> γιατί εμπλέκεται στα τεχνικά πρότυπα διαλειτουργικότητα, αλλά το τέταρτο πακέτο σιδηροδρομικών θεμάτων που μόλι εγκρίνατε θα μα επιτρέψει να ζητήσουμε να τροποποιηθεί όλο το τροχαίο υλικό για την μείωση του θορύβου μέχρι το 2021-2022 όλα τα στοιχεία του τροχαίου υλικού θα έχουν μετασκευαστεί και αυτό θα επιτρέψει στα κάτι μέλη να κάνουν απαραίτητες ενέργειες για την απαγόρευση ορισμένων στοιχείων του τροχαίου υλικού που δεν θα έχουν περάσει αυτή τη μετασκευή στο δικτύο τους. Τέλος κύριε Πρόεδρε, για, τον, για τους κρίκους πρέπει να εξετάσουμε και πάλι την κατάσταση για τα θέματα αυτά. Έχουμε πάρει τη σκητάλη από εσά σε ορισμένα από τα εγχειρήματα που ξεκινήσατε εσείς και λαμβάνουμε υπόψη και αυτά που ζήτησε το Κοινοβούλιο τα προηγούμενα χρόνια. Ελπίζουμε ότι τον Ιούνιο φέτος, στις ημέρες για τα ευρωπαϊκά δίκτυα, θα μπορούμε να σας παρουσιάσουμε κάποια αποτελέσματα για όλα αυτά τα, τους ελείποντες κρίκους που θα έχουμε παρακολουθήσει και εξετάσει και ελπίζω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να στοχεύσουμε καλύτερα σε μια πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για προτάσεις ώστε να καλύψουμε τα κενά και τα χάσματα τα οποία έχουν παραμείνει. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ λέει και ο Πρόεδρος. Έχω και άλλη μια ερώτηση. Τα μεγάλα έργα δεν είναι μόνο το Λιόν Τωρίνο. Υπάρχουν και άλλα τούνελ, παραδείγματο χάρη. Ελέγξατε τι εναλλακτικέ. Γιατί σαφές είναι ότι θα γίνει το Λιόν Αλλά υποτίθεται ότι θα ήταν 12 δις και τώρα μας λένε 26. Και οι χώρες μας λένε πως ε, θα χρηματοδοτηθεί μόνο με 40% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μα άμα είναι έτσι μόνο αυτό θα πληρώσουμε και τίποτα άλλο. Δεν μπορείτε να μας το πείτε, αλλά δεν θα μείνουν άλλα λεφτά. Είχαμε στην ε, Γερμανία την ε, εμπειρία 10 δισεκατομμύρια πήγανε στη Στουτγκάρδη για να γλιτώσουν μερικά λεπτά δρόμο. Συγκεκριμένα λοιπόν ελέγξατε τις εναλλακτικέ. Ή ε, το Λιόν το Ρήνο η φυστάμενη γραμμή. Ή το Ζέμεριγγεν Κόρα. Ήδη ε, μόνο αν ακούσουμε την λέξη της ε, κοιλάδας της Πανωνικής εκεί πέρα αυτό μας λέει, είναι κοιλάδα, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο εύκολο έτσι και είναι πολύ πιο φτηνό και πόσο θα είναι 10 λεπτά πιο αργά θα κάνει κανείς. Πώς μπορείτε λοιπόν να επηρεάσετε την ε, κατάσταση και πώς θα αντιδράσουν τα κράτη-μέλη αν γίνεται τέτοιο. Νομίζω ότι έχουμε εξετάσει όλες τις εναλλακτικέ λύσεις όταν εξετάζαμε τον κανονισμό αυτό σε σχέση και με τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Όλα αυτά όμως είναι ρευστά. Εάν τα σχέδια αυτά εξελίσσονται προς την κατεύθυνση που περιμένουμε, θα εξασφαλίσουμε, θα μπορέσουμε να τα χρηματοδοτήσουμε μέχρι του 40% όπως έχουμε δεσμευτεί και όπως αναφέρεται σαφώς στον κανονισμό. Αν λοιπόν αυτά τα προγράμματα μπορέσουν να προχωρήσουν χωρίς μεγάλα προβλήματα έχει καλώς. Εάν υπάρξουν προβλήματα θα χρειαστεί σε πραγματικό χρόνο να τροποποιήσουμε την χρηματοδότηση και ενδεχομένω να καταλήξουμε και σε διαφορετικά συμπεράσματα. Όλο αυτό το έργο ενορχιστρώνεται μέσα και στο, στα σχέδια εργασίας των διαφόρων συντονιστών. Τα έγγραφα αυτά των συντονιστών θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι γίνονται οι κατάλληλε διαμεσολαβήσει μεταξύ των σχεδίων και τίθενται και οι προτεραιότητε για τη χρηματοδότηση. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι τα σχέδια αυτά εργασία θα παραμείνουν επίκαιρα, θα ενημερώνονται τακτικά και μέσω των εγγράφων αυτών θα έχουμε τη δυνατότητα να τροποποιήσουμε τι πολιτικέ μα εάν παραστεί ανάγκη. Σίγουρα, κύριε Πρόεδρε, αυτή η συζήτηση θα πρέπει να γίνει στο πλήρε πλαίσιο τη προετοιμασία τη επόμενη περίοδου χρηματοδότησης, γιατί θα έχουμε να κάνουμε εκεί και νέες επιλογές σε σχέση με το τι θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε και με τι είδος χρηματοδότησης θέλουμε να καλύψουμε αυτά τα προγράμματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ λοιπόν για τα ερωτήματα και τι απαντήσει. Έχουμε κλείσει το σημείο αυτό τη σημερινή διάταξη και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο τη σημερινή διάταξη, κοινωνικό dumping στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, γνωμοδότηση προς την Επιτροπή ΕΜΠΛ και δίνω το λόγο στον εισηγητή γνωμοδότησης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομος θα είμαι. Θα ήθελα να περιγράψω την κατάσταση πολύ σύντομα. Να σας πω τι λέει η γνωμοδότηση. Αυτή είναι μια γνωμοδότηση που απευθύνεται στην ε, Επιτροπή Επασχόλησης. Έχουμε όμως αποκλειστικές αρμοδιότητες σε κάποιους τομείς και μικτές αρμοδιότητες σε κάποιους ε, άλλους. Και αυτές σε έξι διαφορετικές περιοχές, σε έξι διαφορετικούς τομείς. Σε αυτούς τους έξι τομείς θα επικεντρωθούμε εμείς και θα συζητηθούν και στην Ολομέλεια ούτως ή Είχα δύο συναντήσεις με τους κοιόδης εισηγητές Έχουμε 236 τροπολογίες και προσπαθούμε να τις αποτυπώσουμε σε 18 συμβιβασμούς. Ελπίζω με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε ε, μία τελευταία συνάντηση με τους κοιόδης συζητητές αύριο και να καταλήξουμε. Η αφετηρία μου από την αρχή ήταν, και το έχω πει και κατ' επανάληψη, ότι το θέμα είναι το να εφαρμόσουμε την ισχύουσα νομοθεσία σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό και μόνο αυτό. Επίσης, να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν αποτελεσματικοί έλεγχοι. Πριν περάσω στη γνωμοδότηση και στα επιμέρους σημεία που εμπεριέχονται, που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά, θα ήθελα να σας πω προκαταρτικά ότι στη συζήτηση μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι η το κοινωνικό dumping έχει πολύ διαφορετικές ερμηνείες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην βόρεια Σουηδία, σε μια χώρα όπου προφανώς υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία και κανένα έλεγχο των διαβατηρίων επί 50 χρόνια, τα θέματα των μισθών και τα κοινωνικά θέματα ε, ανάμεσα σε εμά και στην Νορβηγία ε, είναι τελείως διαφορετικά. Παραδείγματο χάρη, είναι πολύ καλύτερα ε, τα πράγματα στην Νορβηγία. Πολλέ νοσοκόμε πήγαν στην Νορβηγία, α πούμε, για να δουλέψουν, γιατί παίρνουν πολύ καλύτερου μισθού. Δηλαδή, ενώ δεν υπάρχει έλεγχο στα σύνορα ανάμεσα στην Σουηδία και στην Νορβηγία, ε, τα πράγματα, οι συνθήκες εργασίας και τα λοιπά στην Νορβηγία είναι πολύ καλύτερες. Επίσης στην πόλη μου ε, συνάντησα έναν αγρονόμο που, είχα, που ήταν έξαλλος γιατί είχε βρει δουλειά στην Ορβηγία και τον ε, υποχρέωσαν όμως να δεχτεί χαμηλότερο μισθό. Σε κάθε χώρα πρέπει να πληρώνεται τουλάχιστον ο ελάχιστος μισθός όμως. Θα πρέπει ο επιχειρηματίας ε, για τον οποίο δούλευε αυτός ο αγρονόμος να πληρώνει τουλάχιστον το βασικό μισθό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το κοινωνικό ντάμπινγκ και ο αθέμητος ανταγωνισμός είναι οι δύο ε, του ίδιου νομίσματος. Θέλουμε να υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός. Θα πρέπει οι συνθήκες ε, που ισχύουν σε μια χώρα, οι συνθήκες ανταγωνισμού, να γίνονται σεβαστές από όλους. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι για τα κοινωνικά θέματα έχουμε εθνικές αρμοδιότητες και τους μισθού. Ε, το κάθε κράτο ε, τους καθορίζει. Έχουμε 28 διαφορετικές πραγματικότητε. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δεχτούμε, να το διαχειριστούμε. Και το κάνουμε με κανόνες Για τις μεταφορές όμως τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί οι μεταφορές ε, αφεαυτών είναι ε, διασυνοριακές. Επομένως, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι πρέπει να εφαρμόσουμε τους κανόνες που ισχύουν τώρα και να ελέγξουμε με αυτόν τον τρόπο την εφαρμογή. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Αλλά επίσης θα πρέπει να παραδεχτώ ότι υπάρχει και κάποια σύνδεση μεταξύ της ε, ασφάλειας για τους επιβάτες και των χρηστών των ε, δρόμων και των κοινωνικών προτύπων και προδιαγραφών. Για μένα είναι σαφής αυτή η σύνδεση. Σε ό,τι τώρα αφορά τα μεμονωμένα σημεία, είναι σωστό να διαπιστώσουμε ότι τα θέματα των ε, οδικών μεταφορών καλύπτονται από πάρα πολλούς κανόνες για το καμποτάζ και άλλα θέματα. Και είναι πολύ δύσκολο να τηρήσουμε όλους αυτούς τους κανόνες. Πάντα μπορεί κανείς να τους παραβιάσει εύκολα, μπορεί να μην υπάρχει αρκετή, αρκετός έλεγχος ή να μην εξασφαλίζεται ότι τηρείται το, τηρούνται οι κανόνες για το καμποτάζ. Αλλά θα πρέπει να απλοποιήσουμε αυτούς τους κανόνες για να είναι πιο δυνατόν, πιο εύκολο να τηρούνται αυτοί οι κανονισμοί και τουλάχιστον να συνομεύονται καλύτερα. Χρειάζεται οπωσδήποτε όμως να υπάρξει εποπτεία της εφαρμογής όλων αυτών των κανόνων. Μία τέτοια μορφή λοιπόν ε, εποπτείας της εφαρμογής των κανόνων θα πρέπει να οργανωθεί από όλους μας, από κοινού. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο σημείο στη γνωμοδότησή μου όπου τονίζω ότι υπάρχει πάντα η δυνατότητα να βελτιώσουμε τους ελέγχους χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και αυτό μπορεί να γίνει στα καινούρια ε, φορτηγά οχήματα με την χρήση της ψηφιοποίησης μπορούμε να έχουμε καλύτερο έλεγχο χωρίς πρόσθετο άχθος πάνω στις εταιρείε μεταφορών. Οι αρχές μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία μπορούν να έχουν καλύτερο έλεγχο της κίνησης των οχημάτων και πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες μας νέα τεχνολογία. Πιστεύω ότι η ψηφιακή τεχνολογία θα διευκολύνει και το έργο των ελεκτικών και εποπτικών αρχών. Είναι επιπλέον απαραίτητο να έχουμε μια στρατηγική που να καλύπτει τις αεροπορικές μεταφορές. Και εδώ θέλω να σας ε, υπενθυμίσω το ότι η σωστή εφαρμογή των συνδικών εργασίας για τις αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να εξασφαλίζεται, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και προηγουμένως κάποια εναρμόνιση και ομοιομορφία των κανόνων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Τι είναι καταρχήν η βάση εργασίας για το υπτάμενο προσωπικό. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να υπόκειται σε ένα ευρωπαϊκό ενιαίο κανονισμό. Και υπάρχουν και τα άλλα θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει στο παρελθόν και πιστεύω Έχω προσπαθήσει να λάβω υπόψη τις διαφορετικές απόψεις των πολιτικών ομάδων και να συγκροτήσω κάποια πλειοψηφία υπέρ αυτής της γνωμοδότησης. Δεν μπορώ βέβαια να περάσω <clears throat> όλα αυτά τα οποία θα ήθελα σε αυτή τη γνωμοδότηση, γιατί υπάρχουν διαφορέ μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Ελπίζω όμως ότι θα μπορέσουμε με τη γνωμοδότηση αυτή να δώσουμε ένα σαφέ μήνυμα προς την Επιτροπή Απασχόληση, λέγοντας ότι για μας ως Επιτροπή Μεταφορών αυτά είναι τα σημαντικά θέματα. Θέλουμε θεμητό ανταγωνισμό, αλλά δεν θέλουμε κοινωνικό dumping. Ευχαριστώ. Ο Μάρκους Πίπα. Ja, Herr Vorsitzender, danke auch an den Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους ε, για την συνεργασία. Πριν από λίγες εβδομάδες συναντηθήκαμε αρκετοί ευρωβουλευτές με διάφορους ε, φορτηγατζίδες που επηρεάζονται από το θέμα το κοινωνικό ντάμπινγκ. Και πρέπει να πω πως ε, η πεμπτουσία ήταν η εξής. Μας ζήτησαν ψηλότερους, ε, ε, σοβαρότερους κανόνες όσον αφορά την παραμονή στο εξωτερικό, το χρόνο οδήγησης και ξεκούρασης. Σωστά όλα αυτά, αλλά το πρόβλημα τελικά καταλήξαμε ότι δεν ήταν οι ελάχιστες προδιαγραφές, αλλά η έλεγχη, η έλεγχη των κρατών μελών η εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Αν δεν λειτουργεί αυτό, θα μπορούμε να βάλουμε εμεί ό,τι προδιαγραφέ θέλουμε. Τα ούτω ή άλλω τζάμπα θα πάνε όλα. Οπότε, να πω κάτι. Ε, δεν εκμεταλλεύονται όλες οι επιχειρήσεις τους οδηγού. Υπάρχουν εξαιρετικά παραδείγματα που λειτουργούν υποδειγματικά συνεργάζονται με τα συνδικάτα, με τους οδηγούς. Έχουν πάρα πολύ καλά κοινωνικά μοντέλα. Δεν μπορεί να τα βάζουμε όλα σε ένα κουβά. Αλλά γεγονός είναι ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και επειδή υπάρχει ευρωπαϊκή διάσταση, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές ιδέες. Για τη γνωμοδότηση τώρα την ίδια. Πρώτα απ' όλα χαιρετίζουμε το ότι η Επιτροπή ε, Μεταφορών επιμένει ότι είναι δική της ε, αρμοδιότητα, δεν μπορεί να μπαίνει εδώ πέρα η Επιτροπή Απασχόλησης. Εδώ συμφωνούμε με τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, και τον εισηγητή. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν αυτά τα πράγματα. Όσον αφορά το συγκεκριμένο περιεχόμενο, να ξαναπώ πως από την αρχική πρόταση του εισηγητή είχαμε πολλά πράγματα τα οποία είπαμε στις συμβαστικές προτάσεις και μάλλον τελικά θα έχουμε μια καλή γνωμοδότηση με μεγάλη πλειοψηφία. Έχουμε 18 συμβαστικές προτάσεις, 9 τις λάβαμε μόλις χτες. Θα πρέπει να συνοηθούμε. Αλλά για εμάς είναι σαφές ότι νέες αρμοδιότητες ελέγχου της Κομισιόν δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν και δεν πρέπει να είναι στην έκθεση άρα. Γιατί αυτό θα δημιουργήσει λανθασμένες προσδοκίες που δεν έχουν, δεν μπορούν να γίνουν με τις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες. Θα ζητήσουμε λοιπόν την αρχή της επικουρικότητας. Τα κράτη-μέλη πρέπει να ελέγχουν και να εφαρμόζουν. και η Κομισιόν μπορεί να συντονίζει εδώ πέρα. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει να βρει τα προβληματικά θέματα. Οπωσδήποτε λοιπόν ναι, ο ρόλος ο συντονιστικός είναι σημαντικός. Και προς αυτή την κατεύθυνση επίσης είναι το ότι δεν χρειαζόμαστε πάλι νέα ευρωπαϊκή υπηρεσία για τους αυτοκινητοδρόμους. Δεν είναι προς συζήτηση, δεν είναι αυτό το θέμα, μπορούμε να το δούμε αργότερα. Αλλά δεν μπορεί, δεν έχει σχέση τώρα με το κοινωνικό ντάμπινγκ να πούμε να φτιάξουμε νέα υπηρεσία. Με κολλάει εδώ. Επίσης, θετικό το ότι διαγράφηκε και η απέτηση η οποία ζητούσε πάλι ένα νέο κανονισμό. Όλα τα άλλα νομίζω κύριε Νίλσεν θα μπορέσουμε να τα δούμε στους συμβιβασμούς. Και προσωπικά έχω κάθε καλή διάθεση για να έχουμε μια σωστή γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ Ρόμπερτ Σίλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Γιάννη Νίλσεν. Η διαδικασία ήταν πάρα πολύ δημοκρατική. Είχαμε δύο συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών. Από αυτή την σκοπιά δεν έχω κανένα παράπονο. Και μετά τον τελευταίο γύρο συναντήσεων με τους σκιώδεις εισηγητές ε, υπήρξε βελτίωση όπως η συμβαστική λύση 4 που υπάρχει σύνδεση με τα προστατευτικά μέτρα που χρησιμοποιούνται σε ορισμένε περιπτώσεις εντελώς αδικαιολόγητα. Όμως Πρέπει να πω ότι και μετά από αυτές τις συναντήσεις, διαπραγματεύσεις και τα λοιπά με τους Κιώδης, ξεφεύγουμε από την ιδεολογία της ε, Επιτροπής Μεταφορών και στερνιζόμαστε την ε, ιδεολογία της Επιτροπής Απασχόλησης. Ε, η κατάσταση στην, στους συνδροδρόμους, στους αυτοκινητοδρόμους, στις εναέριες κυκλοφορίες στην ναι, αεραία κυκλοφορία και, στις, και στο λιμάν, στα λιμάνια είναι τελείω διαφορετικέ και μερικέ φορέ θα αντιμετωπίσουμε σαν το ίδιο πράγμα. Παραδείγματο χάρη, οι νέοι και οι γυναίκε θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να μπουν στι στις μεταφορές. Ε, καλή ιδέα, αλλά για πολλούς νέους άνεργους σε διαφορετικές χώρες ε, είναι τελείως διαφορετικές οι προϋποθέσεις για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Παραδείγματος χάρη στις μεσογειακές χώρες έχουμε πολύ ψηλή ανεργία των νέων. Ε, και αν θέλουμε να βάλουμε τέτοιες φράσεις ε, στο κείμενό μας, θα πρέπει να μιλήσουμε και για τα εμπόδια τα οποία, στα οποία προσκρούν οι νέοι και δεν μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Επομένως, θα πρέπει να αρθούν αυτά τα εμπόδια, άρα θα πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία. Ε, στους συμβιβασμούς 6 και 7 υπάρχει αυτή η ιδέα εξάλληψης κάποιων επιχειρήσεων, εξαφάνισης ας πούμε κάποιων επιχειρήσεων από τις ε, επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δηλαδή ένα είδος ε, μαυροπίνακα ας πούμε, που γράφονται οι επιχειρήσεις ας πούμε. Δεν είναι καλή ιδέα αυτή. Παραδείγματο χάρη ε, έχουμε κάποιες παράνομες εταιρείε στην στις χερσαίες μεταφορές και έχουμε και τα και τις σημαίες ευκαιρίας που είναι κάτι τελείως ε, νόμιμο. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Επίσης, οι, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, λέμε, μιας ε, επιχείρησης ε, σε, σε μια, στην αγορά μιας χώρας στην οποία δεν είναι εγκατεστημένη θα είναι εντελώς προσωρινές. Πηγαίνουμε σε τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις. Επίσης, ε, αυτό το παράδειγμα που δώσατε για την ε, Βόρεια Θάλασσα και την Νορβηγία είναι σωστό. Είναι λογικό όμως, ας πούμε, κάποιες επιχειρήσεις να, έρχονται να μπαίνουν σε κάποιες ε, αγορές και τους συμφέρει. Αν τώρα ε, χρησιμοποιήσω τις ε, υπηρεσίες ενός ε, κράτους για να κάνω κοινωνικό dumping, αυτό δεν είναι καλό. Αλλά αν πραγματικά κάνω, πηγαίνω σε μια ξένη χώρα και κάνω την ίδια δουλειά, ας πούμε, σε αυτή τη χώρα, με, σεβόμενος τους κανόνες της χώρας ε, αυτής, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και δεν πρέπει να υπάρχει καμία διακριτική μεταχείριση σε αυτήν την περίπτωση. Όταν μιλάμε για κοινωνικό ε, dumping, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε εδώ μια ενία αγορά και στις μεταφορές έχουμε μια ενία αγορά και μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο μας η ενία αγορά. Τελέσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νίλσον και εγώ συμφωνώ για το γεγονός ότι είχαμε πολύ ανοιχτέ συζητήσεις και ο με τον εισηγητή. Ο εισηγητή ήταν ιδιαίτερα διατεθειμένο να δεχτεί και τι προτάσει των σκιωδών. Προφανώ θα υπάρξουν τελικά διαφορέ απόψεων για μεμονωμένα σημεία και ο εισηγητή έχει κάθε δικαίωμα ενδεχομένω να μην λάβει υπόψη τι προτάσει των σκιωδών εάν εάν δεν συν, συνάδουν με τη γενική του κατεύθυνση. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Νίλσεν και να υποστηρίξω αυτά που είπε ότι πρέπει να έχουμε μια ευρεία πλειοψηφία ως Επιτροπή Μεταφορών για το θέμα αυτό <clears throat> και κατανοεί ότι έχουμε ακόμα κάποιο δρόμο να διαθέξουμε. Να σταθώ σε μερικά πιο ουσιαστικά σημεία. Για τις λεπτομέρειες θα συναντηθούν και πάλι οι σκιώδεις εισηγητές αύριο και γι' αυτό ίσως είναι καλύτερα να τα δούμε στις συνεδρίες των, των ε, σκιωδών. Πρώτα απ' όλα, δεν θεωρώ ότι έχουμε τη σωστή ισορροπία ακόμα μεταξύ της πτυχής της κοινωνικής και της πτυχής απασχόλησης και της πτυχής της αγοράς. Έχουμε το στόχο αυτό, υπάρχει και στη φρασιολογία, θέλουμε να έχουμε θεμητό ανταγωνισμό χωρίς κοινωνικό ντάμπινγκ, αλλά αν δούμε πιο προσεκτικά τα θέματα θα συμφωνήσω με τον Προλαλήσαντα που είπε ότι δεν έχουμε προχωρήσει λιγάκι προ την κατεύθυνση τη Επιτροπή Απασχόληση και δεν έχουμε κρατήσει τη σαφή γραμμή τη επιτροπή Μεταφορών. Αυτό λοιπόν πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε καλύτερα. Επίση, κανεί από εμά δεν θέλει το κοινωνικό ντάμπινγκ. Αυτό είναι σαφέ, Όπω είπε και ο κύριο Νίλσεν όμω, υπάρχουν διαφορετικέ αντιλήψει και διαφορετικοί ορισμοί για το κοινωνικό ντάμπινγκ και εκεί πρέπει να εστιάσουμε αύριο το, στη συνάντηση των σκιωδών να κατανοήσουμε όλοι ότι μιλάμε όλοι για το κοινωνικό ντάμπινγκ και όχι για διαφορετικούς στόχους και διαφορετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα. Γιατί και αυτά είναι ένα κομμάτι της προβληματικής της εσωτερικής αγοράς. Το τρίτο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι σε κάποιες από τις ε, παραγράφους, και το είπε ο Ρόμπερτ Σίλα, εμείς ξεπερνάμε τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και αυτά που αναφέρονται στη συμβαστική τροπολογία 6. Εκεί που ζητάμε την Κομισιόν να διερευνήσει το κοινωνικό ντάμπινγκ σε όλους τους τομείς μεταφορών και να εφαρμόσει κυρώσεις σε εταιρείες που παραδιάζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες κτλ. κτλ. Εδώ αναμειγνύουμε λιγάκι θέματα αρμοδιοτήτων των κρατών μελών αφενός και της Κομισιόν αφετέρου. Αυτό για μένα είναι το πιο προβληματικό ε, στοιχείο μεταξύ, μεταξύ των τροπολογιών συμβιβασμού. Και θα ήθελα λοιπόν να το τροποποιήσουμε λιγάκι εκεί ως προς τη διατύπωση. Και βλέπω ότι και οι σιώδεις ηγητές είναι κάπως διχασμένοι για το θέμα αυτό. Θα είναι δύσκολο να έχουμε μια πλειοψηφία, αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία μπορούμε να διατηρήσουμε. Μιλάμε για το κοινωνικό dumping. Όταν το λέμε αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι όλοι θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες συνθήκες εργασίας και αποδοχές. Συμφωνήσαμε με τον κύριο Νίρσε στην τελευταία ε, συνεδρίασή μας, συνάντησή μας ότι μιλάμε για ισότητα ανταγωνισμού και συγχρόνως ισότητα ευκαιριών. Και αυτό πρέπει να διατρέχει όλο το κείμενο. Χωρίς όμως να δείξει την ποιότητα του, της γνωμοδότησής μας. Θα σταματήσω εδώ γιατί νομίζω ότι κάποια άλλα θέματα για τα οποία θα ήθελα να αναφερθώ είναι εν γνώση μόνο των σκιωδών και όχι των υπολείπων μελών της Επιτροπής. Δεν είμαστε μακριά από το τελικό νήμα. Έχουμε κάποιες ε, ε τροπολογίες συμβασμού που μπορεί να είναι αμφιλεγόμενες και έχουμε κάποια σημεία που πρέπει να τροποποιήσουμε και να βελτιώσουμε την ε, διατύπωση, αλλά έχω κάθε ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα μπορέσει να υποστηριχθεί από μια ευρεία πλειοψηφία αύριο. Ευχαριστώ. Η Κατερίνα Κονέτσινα. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για την γνωμοδότηση. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να γράψει κανείς μια γνωμοδότηση για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα και δεδομένη της κατάστασης στο Κοινοβούλιο και να βρει μια λύση στις τροπολογίες. Αλλά θα αρνηθείτε τη σχετικοποίηση του προβλήματος και θα υποστηρίξετε με νύχια και με δόντια το κείμενο που γράψατε. Γιατί έχουμε χώρο μόνο για γεγονότα σε ένα τέτοιο κείμενο. Και εγώ πιστεύω, όπως και εσείς, ότι η ασφάλεια των επιβατών και οι συνθήκες εργασίας ε, θα πρέπει να ενσωματωθούν στη λογική του τομέα των μεταφορών. Και λέξεις ε, όπως το θνητικό μέι, στο κείμενο είναι πάρα πολύ αρνητικές. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής ε, ισότητα ε, και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να διακυβεύεται η ασφάλεια στον τομέα των μεταφορών. Συμφωνώ με πάρα πολλέ από τι τροπολογίε και του συμβιβασμού, αλλά σα προειδοποιώ να μην είμαστε αφελεί και απλουστευτικοί. Το 2014, 1,9 εκατομμύρια εργαζόμενοι πήγαν στο εξωτερικό και συχνά ε, πολλοί από αυτούς εργάστηκαν ε, στον τομέα των μεταφορών. Ήταν ε, μία αύξηση του 10%. Συχνά ο εργοδότης τους του ζήτησε να πάει να δουλέψει στο εξωτερικό και θα έπρεπε να πάρουν τον ίδιο μισθό με τους ντόπιου. Εάν ε, δουλεύεις σε μια ξένη χώρα και κάνεις την ίδια δουλειά με τον γηγενή αλλά πληρώνεις διαφορετικά, δεν είναι δίκαιο αυτό. Θα πρέπει ε, και ο αποσπασμένος εργαζόμενος να πληρώνεται τα ίδια με τον γηγενή. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πούμε από την άλλη βέβαια ότι οποιαδήποτε διαφορά στους μισθούς αυτόματα είναι κοινωνικό dumping, αλλά το να προσπαθούμε εν ονόματι τη ανταγωνιστικότητα να κρατάμε στον πιο χαμηλά του μισθού, αυτό είναι κατά των αρχών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι που θέλετε να εισαχθούν τεχνολογίε ούτω ώστε να βελτιωθούν οι έλεγχοι στον τομέα των μεταφορών, ε, να παρακολουθούμε τον χρόνο εργασίας ε, των εργαζομένων, να εξασφαλίσουμε ότι η ισχύουσα νομοθεσία εφαρμόζεται. Όλα αυτά είναι τέλεια, τα υποστηρίζω. Επίσης, όλοι θέλουμε να έχουμε οδηγούς οι οποίοι είναι ξεκούραστοι, γιατί αυτό είναι προς το συμφέρον της ασφάλειας στους ε, δρόμους και η ασφάλεια στους δρόμους και η επαρκής ανάπαυση των οδηγών είναι ε, πράγματα που συνδέονται πάρα πολύ. Θέλω να κρατήσουμε όλες τις θετικές ε, απόψεις που υπάρχουν στη γνωμοδότηση. Ντέλη, η κυρία Ντέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για τις προτάσεις και τις συμβαστικές προτάσεις. Εγώ θα ήθελα να σε επιθέσω την προσοχή σε ένα γεγονός. Ακόμα και αν ο κύριος Γιούνκερ θεωρεί ότι είναι η Επιτροπή της τελευταίας ευκαιρίας αυτή, δεν μπορούμε να τα κάνουμε μαντάρα στο θέμα του κοινωνικού ντάμπινγκ. Γιατί είτε το πούμε κοινωνικό ντάμπινγκ είτε εκμετάλλευση των εργαζομένων το ίδιο κάνει. Είναι το δηλητήριο που σκοτώνει την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Όλο και περισσότερο βλέπουμε ότι τελικά δεν γίνεται τίποτα γύρω από αυτό το θέμα και τελικά οι πολίτες μας δεν έχουν την εμπιστοσύνη στην Ευρώπη που θα έπρεπε να έχουν, γιατί η Ευρώπη στο μυαλό τους θα πρέπει να τους προστατεύσει, θα πρέπει να προστατεύει και τους εργαζόμενους και δεν το κάνει. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι η κατάσταση είναι καταστροφική. Ειδικά όταν βλέπετε τους μισθούς, γίνεται μια κούρσα προς τα κάτω. Επίσης, το θέμα της ασφάλειας και της ε, υγείας ε, στο χώρο εργασίας είναι σκανδαλώδη. Ε, οι συνθήκες μερικές φορές είναι σκανδαλώδεις. Καταστροφικές και αναξιοπρεπείς. Και επίσης, υπάρχει ένα φαινόμενο όπου κάποιοι οδηγοί φορτηγών υφίστανται συνεχή πίεση, ορισμένοι υποχρεούνται από τους εργοδότες τους να ξεκουραστούν μέσα στο φορτηγό τους, επί εβδομάδες, μέσα σε συνθήκες απαράδεκτες. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε λίγο κουράγιο να τα πούμε τα πράγματα. Ακούω συναδέλφους που λένε ναι, αλλά εξαρτάται από το ένα και το, το άλλο, από την νομοθεσία των κρατών μελών και ο κ. Ζήλερ μίλησε για τους μισθούς των ευρωβουλευτών. Έτσι, έχουμε όλοι τον ίδιο μισθό. Γιατί γιατί ακριβώς θέλαμε να προβάλλουμε αυτή την ιδέα της, των εναρμονισμένων μισθών. Παλιά ο Ιταλός έπαιρνε το μισθό του Ιταλού ε, βουλευτή, ο Γερμανός του Γερμανού, τώρα όλοι το ίδιο. Αυτό τι, με αυτό τι θέλω να πω, ότι χρειαζόμαστε κάποια ελάχιστα, ένα κατόφλι, κάποια ελάχιστα στους μισθούς, κάποια ελάχιστα όρια. Και στους μισθούς, αλλά και στις συνθήκες εργασίας. Αυτά τα ελάχιστα όρια θα πρέπει να τα εξασφαλίσουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μετά. Έπειτα. Πώς Το μήλο της έρηδος είναι το θέμα των ελέγχων. Θα πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σώμα επιθεωρητών το οποίο ελέγχει ακριβώς θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες οι οποίοι γίνονται ε, σεβαστοί, θα πρέπει να εφαρμοστούν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χρειαζόμαστε λιγότερους κανόνες, όχι. Τους χρειαζόμαστε τους κανόνες και να τους ελέγχουμε. Επίσης, θα πρέπει να εξαλείψουμε την ψεύτο ε, υπερκολαβία. Ορισμένοι συνάδελφοι λένε, όχι δεν συμφωνώ να, βάλουμε, να φτιάξουμε ένα μαυροπίνακα. Μα έχουμε και μαυροπίνακα με αεροπορικές εταιρείε που δεν ε, λειτουργούν σωστά. Γιατί θα έχουμε αυτό το μαύρο πίνακα, για να επιβραβεύσουμε αυτούς που σέβονται τους κανόνες και για να στυλιτεύσουμε τους υπόλοιπους. Και θα πρέπει οι εταιρείε να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ο κύριος Ζήλερ επίσης είπε κάτι πολύ σωστό. Όταν μιλάμε για τις μεταφορές και ο εναέριος τομέας, βλέπετε τι γίνεται με τη Ryanair, βλέπετε τι γίνεται στις χερσαίες μεταφορές, αλλά και στις θαλάσσιες μεταφορές υπάρχει μια εκμετάλλευση των, ε, των εργαζομένων, ε, μοντέρνα εκμετάλλευση με αδήλωτους εργαζόμενους που είναι παράδεκτη. Στην αυριανή ε, συνεδρίαση ελπίζω το αποτέλεσμα να είναι θετικό. Θα πρέπει η Ευρώπη να πάει προς τα εμπρός. Θα πρέπει να υπάρξει μια γνωμοδότηση που οι πολίτες θα, όταν τη διαβάσουν θα δουν ότι εμείς τους υπερασπιζόμαστε. Σήμερα πρέπει να ρυθμίσουμε αυτά τα πράγματα, όχι αύριο μεθαύριο. Είτε θα μιλήσουμε για μια Ευρώπη που προστατεύει, είτε θα προβάλλουμε την εικόνα μιας Ευρώπης που καταστρέφει και θα, χάθουν, θα χαθεί για πάντα η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών σε αυτήν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την δουλειά που έχετε κάνει με τη γνωμοδότηση αυτή και για τις ε, συζητήσεις που κάνουμε. Θα ήθελα να πω πως βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Είτε θέλουμε δηλαδή σωστούς κανόνες και καλές συνθήκες εργασίας ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή μέχρι τώρα λέμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες, είναι ένας ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών. Θεωρώ πως εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε συμμετοχή σε εκλογές κάτω από 50%, οι τόνοι έχουν οξυνθεί στη δε χώρα μου, στη Σουηδία. Μπορώ να σας πω πως η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ χαμηλή. Ελπίζω πραγματικά να προχωρήσουμε όσον αφορά το καμποτάζ και τον έλεγχο των κανόνων γιατί υπάρχουν θέματα κοινωνικού ντάμπινγκ στον τομέα των μεταφορών. Ο τομέας αυτός αλλάζει, πρέπει να μπουν νέοι στον κλάδο να είναι ελκυστικός, αλλά όπως έχουν τώρα τα πράγματα, αλλά θα πρέπει κάποιος να μπορεί να ζει και να ζει στην οικογένειά του από, αυτό το, από αυτή τη δουλειά. Αλλιώ δεν γίνεται έτσι, να μην μιλήσω για τις συνθήκε στις οποίες ζουν, το να μην βρίσκουν ένα πάρκινγκ ε, στην άκρη του αυτοκινητοδρόμου, δεν είναι ελκυστικέ συνθήκε αυτές για τους ε, νέους. Πρέπει λοιπόν να είμαστε υπέρ ενό δικαίου ανταγωνισμού. Επίσης διαπιστώνω συχνά στην συζήτηση πως στα λεγόμενα παλιά κράτη-μέλη η κατάσταση είναι εξής. Έχουμε νέους οδηγούς που έρχονται από τα παλιά κράτη-μέλη και εντείνουν τον ανταγωνισμό γιατί είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν με τα μισά λεφτά. Και αυτό ακριβώς σημαίνει στη χώρα μου οι αλλοδαποί εργαζόμενοι προσπαθούν να μπουν στην αγορά της ε, Σουηδίας θα πρέπει να τηρούν ε, τους νόμους και τους κανόνες. Παρ' όλα αυτά τα σύνορα είναι ανοιχτά, οπότε ο κανονισμός είναι αυτός που περιέγραψα. Οπότε ήθελα να σας πω πως έχουμε, βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει να υπάρχουν σωστές συνθήκες εργασίας ε, και ζωής για όσους δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Αλλιώ απομακρυνόμαστε όλο και περισσότερο από το να εμπιστεύονται οι πολίτες στην Ένωση. Ευχαριστώ. Σεύσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλό είναι που συζητάμε για το κοινωνικό dumping. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα όμως σε όλους, αλλά προηγουμένως να σταθώ ιδιαίτερα. Να ζητήσω από την Κομισιόν να μου, να μου εξηγήσει τι είναι το κοινωνικό dumping. Κάθε φορά που διαβάζω για το κοινωνικό dumping δεν υπάρχει πουθενά ένα ορισμό. Γιατί μιλάμε λοιπόν, αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο που πρέπει να διευκρινίσουμε. Άμα δεν υπάρχει ορισμός είναι μια καθαρά υποκειμενική εκτίμηση τη κατάσταση από τον καθένα και μπορεί ορισμένοι να το χρησιμοποιούν ως ένα πρόσχημα για να εξαλείψουν τον ανταγωνισμό που είναι μια από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Αν λοιπόν έχουμε εταιρείε οι οποίες λειτουργούν σε μια χώρα και θέλουν να διαλέξουν την πιο φθηνή υπηρεσία, θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν αυτή την εταιρεία κάποιοι άλλοι θα πούν «Α, όχι, αυτό είναι κοινωνικό ντάμπινγκ». Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορούν να δοκιμήσουμε αν δεν έχουμε εξασφαλίσει ένα κοινό ορισμό του τι είναι το κοινωνικό ντάμπινγκ. Όταν εγώ κατεβαίνω στο, στην κατίνα του Κοινοβουλίου, βλέπω να υπάρχει διαφορετική τιμή, παραγωγή χάρη για τα μήλα και τα αχλάδια που έρχονται από διαφορετικές χώρες. Μα εκεί υπάρχουν διαφορετικά διαφορετικό κόστος παραγωγής, διαφορετικό κόστος ε, μεταφοράς κτλ. Πώς καταλήγουν να έχουν την ίδια τιμή. Καταλαβαίνω αυτούς που λένε ότι πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν εταιρείε απλώς γραμματοκιβωτίου που εκμεταλλεύονται οδηγούς από την Ανατολική Ευρώπη. Και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο συζητούμε εμείς για το δύσκολο αυτό θέμα σήμερα. Είπατε ότι οργανώσατε μία συνάντηση με οδηγούς φορτηγών είπαν ότι τους εκμεταλλεύονται, αλλά δεν τους εκμεταλλεύονται στις δικές τους χώρες. Είναι δυτικοευρωπαϊκές εταιρείες που τους εκμεταλλεύονται, τους βάζουν να οδηγούν αλλού και τους βάζουν του να δουλεύουν με βουλγαρικούς ή ρουμανικούς μισθούς ενώ δουλεύουν στη Δυτική Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τον αγώνα κατά κάθε μορφής κατάχρησης και εκμετάλλευσης και να εξασφαλίσουμε ότι θα εφαρμόσει η νομοθεσία. Γιατί η επιθεωρήση για τα θέματα αυτά είναι απαραίτητο να γίνονται σε όλες τις χώρες, το απαιτεί η νομοθεσία, αλλά υπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος διαφορετικές ρυθμίσεις για το χρόνο εργασίας και για τις αμοιβέ. Άλλοι πληρώνονται με το μήνα όπως στην Πολωνία, άλλοι πληρώνονται με την ώρα. Δεν θέλω λοιπόν να υποτιμήσω το έργο του εισηγητή, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή εργασία όπως και όλοι οι σκιώδες. Ξέρω ότι είναι δύσκολο το έργο του. Δεν θέλω να υποτιμήσω αυτά που κάνει. Καταλαβαίνω τα σχόλια που έχουν διατυπωθεί από τους διάφορους ε, βουλευτές που προέρχονται από άλλες χώρες. Ξέρω ότι υπάρχει πολλές φορές πίεση η οποία ασκείται από τις μεταφορικές εταιρείες γιατί κινδυνεύουν να χάσουν μερίδια αγοράς από άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν διαφορετική πολιτική ε, αμοιβών. Και φυσικά η φορολογία δεν είναι πάντα η ίδια. Είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα και δεν μπορούμε να έχουμε μια εναρμόνιση μόνο με τον κατώτερο κοινό παρανομαστή. Αλλά εφόσον εδώ η Κομισιόν παρούσα, θέλω να σα ρωτήσω ποιο είναι ο ορισμό του κοινωνικού ντάμπινγκ, αλλά και δύο περαιτέρω ερωτήματα θέλω να θέσω στην Κομισιόν. Πρώτη η Κομισιόν να υπάρξει μια αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων. Αυτό αφήνει ανοιχτό το θέμα του κατά πόσο αυτή η μεταρρύθμιση θα εστιάσει και στους εργαζόμενους στις μεταφορές και ιδίως αυτούς που ασκούν το καμποτάζ. Μπορεί να μας εξηγήσει τώρα η Κομισιόν ποιο θα είναι το καθεστώς των οδηγών φορτηγατζίδων όταν εκτελούν διαμεθοριακές μεταφορές. Επίσης, Ο κανονισμός 561 του 2006 προτείνεται να αλλάξει και αυτός κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να επιτρέπεται στους ε, οδηγούς να ανακτούν τον χρόνο να έχουν τη δυνατότητα ένα, αυτό, ένα μέρος του χρόνου αναπαυσής τους να τον έχουν στην χώρα προέλευσής τους. Η Κριστίν Ρεβουντάλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι είναι προβληματικό το κοινωνικό ντάμπινγκ εναντί των εργαζομένων, εναντί της ε, κοινωνικής τάξης στην Ευρώπη. Έχει επιπτώσεις και στην ασφάλεια, ανησυχεί πολλούς πολίτες μας και πολλούς βουλευτές της Επιτροπής μας και αυτό φάνηκε και από το μεγάλο αριθμό των τροπολογιών που έχουν κατατέθει. Εγώ θέλω να χαιρετήσω το έργο του Γιένς Νίλσεν και των συνεισηγητών τους για το θέμα αυτό, ακόμα και δεν έχουν περατωθεί οι συζητήσεις. Έχουμε 18 τροπολογίες συμβασμού και ευχαριστώ τον Γιένς για την εργασία που έφερε σε πέρα. Τα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά την ε, περασμένη Παρασκευή στη Γαλλία έλαβε χώρα μια δικαστική απόφαση με το δικαστήριο της ε, Βαρένης σε σχέση με έξι μεταφορές, μεταφορείς. Του ζήτησε έξι έτη φυλάξης με αναστολή και πρόστιμο γιατί είχαν ε, απασχολήσει παρανόμως ε, Πορτογάλους, Ρουμάνους και Πολωνούς εργαζομένους πληρώνοντάς τους τις ταρίφες της χώρας τους ενώ δουλεύανε στην Γαλλία. Αυτή λοιπόν είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης στη Γαλλία και βλέπουμε σήμερα ότι η εφαρμογή των κανονισμών και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εξασφαλίσετε η σωστή εφαρμογή τους. Και γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να αφαιθούμε στην στάση των κρατών μελών. Δεν φτάνει κάτι τέτοιο όμως και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός φορέας ο οποίος θα είναι αρμόδιος. αυτά ξέρω ότι η Κομισιόν δεν, δημιουργεί, δεν θέλει να δημιουργήσει νέους φορείς επειδή υπάρχουν προβλήματα στενότητας του προπολογισμού. Αλλά θα μπορούσαμε να φανταστούμε ω ιδρομικός φορέας για τον οποίο εμείς ψηφίσαμε πριν από λίγες ώρες να μπορέσει να γίνει ένα ευρύτερο φορέα για όλε τι χερσαίε μεταφορέ, οπότε να περιλαμβάνει και τι οδικέ μεταφορές και επομένω με τον τρόπο αυτό μπορούμε <clears throat> να εξασφαλίσουμε ότι τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και του σεβασμού των κανόνων ανάπαυση για του οδηγού και για τις, οι κανόνες για τις μεταφορικές εταιρείε, όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν από αυτό το φορέα χωρίς να δημιουργηθεί και ένας περαιτέρω νέος φορέας αλλά να υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών και επιβολή κυρώσεων εναντίον αυτών οι οποίοι δεν σέβονται την κείμενη νομοθεσία. Χαίρομαι λοιπόν γιατί υπάρχουν ορισμένε τροπολογίε που εγώ είχα προτείνει και οι οποίε περιλήφθηκαν στι τροπολογίε συμβιβασμού, άλλε όμω όχι. Δεν ξέρω τι. Ξέρω ότι δεν μπορούν όλα να συμπεριλαμβάνονται στι τροπολογίε συμβιβασμού, αλλά έχουμε την κοινή θέληση να εξασφαλίσουμε ότι στο τέλο αυτή τη συζήτηση που συνεχίζεται φυσικά και προχωρά να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που θα αποτελεί τη γνωμοδότηση τη Επιτροπή Μεταφορών που θα είναι ιδιαίτερα στεναρή για τα θέματα αυτά, γιατί όλοι ανησυχούμε για τα ζητήματα αυτά. Ευχαριστώ. Ο Πίτερ Φαντάρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, Είμαι έξι χρόνια βουλευτής ε, και κάθε χρόνο έχουμε συναντήσεις για κοινωνικό ντάμπινγκ και μιλάμε για οδηγούς, πιλότους, ε, ναυτικούς ε, και την τελευταία φορά ήμασταν στο Ρότερνταμ τον Νοέμβριο με τον συνάδελφο Διγιών από το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και σε όλες αυτές τις συναντήσεις κύριε Πρόεδρε υπάρχει μια κοινή γραμμή και είμαι κάθε φορά περίεργος να δω το τι θα συμβεί. Φοβάμαι ότι υπάρχει πάρα πολύ ιδεολογικοποίηση της ε, συζήτησης, αλλά δεν ε, χρειαζόμαστε αυτό. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι μια πρακτική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Και δεύτερον, αυτοί που λένε «Α, να, θα ξαναφτιάξουμε άλλη μια υπηρεσία εδώ πέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ε, έχω να πω μόνο «Μην το κάνετε». Πρέπει να έχουμε κάποιες απλές πρακτικές επιλογές. Ας ξεκινήσουμε από τον ορισμό του κοινωνικού ντάμπινγκ. Αυτό σημαίνει κοινωνικό ντάμπινγκ ότι έχουμε κάποιες ε, εταιρείε οι οποίες ε, κατ' ουσίαν είναι μόνο γραμματοκιβώτια και με αυτόν τον τρόπο παρακάμπτουν τους ε, κανόνες υπέρ των εργαζομένων. Τόσο απλό είναι, δεν ανάγκη να ανακατεύουμε άσχετα πράγματα. Το χαρακτηριστικό είναι να έχουμε εταιρείες, ε, ε, γραμματοκιβώτια που εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους. Πρώτον. Δεύτερον, σωστά αναφέρθηκε η ασφάλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό φαινόμενο. Βλέπετε πως η οδηγοί αναγκάζονται να ξεπερνούν το χρόνο οδήγησης και εξεκούρασης, αλλά και για τους ε, εργοδότες είναι καμιά φορά φτηνότερο να πληρώνουν τα πρόστιμα από το να σέβονται την νομοθεσία. Και τρίτον, καταπολέμηση της απάτης. Ε, έχετε και εδώ πέρα, αλλά η καλύτερη καταπολέμηση της ε, απάτης γίνεται μέσω της εφορίας. βλέπετε πως εταιρείε που εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους αντιμετωπίζονται καλύτερα μέσω φορολογικών διαδικασιών, μέσω των φορολογικών ελέγχων. Εγώ όταν ήμουν διευθυντής ε, σε μια τέτοια υπηρεσία, ακριβώς για την ε, ναυτιλία συγκεκριμένα, ακριβώς αυτό κάναμε. γιατί εγώ ζήτησα διευκρινήσεις ε, από την Επίτροπο και μου έδωσε μια απάντηση που δεν έλεγε τίποτα, αλλά ας ξεχάσουμε την Κομισιόν. Οι εθνικές υπηρεσίες ελέγχου πρέπει να ασκήσουν πίεση και να πάρουν στα σοβαρά αυτή την υπόθεση. Και βεβαίως το θέμα είναι και η πρόληψη Πρόληψη όμως σημαίνει και κατάλληλα πάρκινγκ στους ε, αυτοκινητοδρόμους να μπορούν να ξεκουράζονται οι άνθρωποι και πάρα πολύ σημαντικό ο έλεγχος. Ο έλεγχος, ναι, εναρμόνιση των ελέγχων Υπάρχει επίσης ε, και μία υπηρεσία σχετική που λέγεται Eurocontrol Route ε, που, στο Λουξεμβούργο που μπορεί κανείς να κάνει ε, ανώνυμες καταγγελίες προς τις ελεκτικές αρχές. Και υπάρχει εκεί βάση δεδομένων αυτών. Οπότε ας αφήσουμε την Κομισιόν δεν ανάγκη να φτιάξουμε και άλλη υπηρεσία. Βλέπετε ότι τα θέματα αυτά πρέπει να λυθούν στην πράξη. Αυτά για να απομακρυνθούμε λίγο από την ιδεολογία και τις φιλοσοφία να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα αυτά τα οποία έχουμε για να καταπολεμήσουμε αυτές τις εταιρείε γραμματοκιβώτια που υπάρχουν και στην εσωτερική ναυσιπλοεία και στην αεροπορία και Ευχαριστώ. Δίτερ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ βεβαίως ε, και τον εισηγητή. Να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Ε, πάντα συναντήσεις με εργαζόμενους ε, μας λένε πως οι επιχειρήσεις εξωθούν τους εργαζόμενους να παραβιάσουν τους κανόνες και προτιμούν να πληρώνουν τα πρόστιμα γιατί είναι φθηνότερο. Οπότε στο... στην τροπολογία 29 ζητάω ακριβώς να υπάρχουν ποινές και πρόστιμα με αποτρεπτικό χαρακτήρα. Δεύτερον, έχουμε πάρα πολλά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από τα ηλεκτρονικά διόδια, αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό προτείνω στην τροπολογία 103 οι αρχές να έχουν πρόσβαση τα δεδομένα των ηλεκτρονικών διοδίων για να ελέγχουν καλύτερα τις απαιτήσει για το καμποτάζ. Ο συνάδελφος μόλις μίλησε για πρακτικές λύσεις, νομίζω αυτή είναι μια πρακτική λύση. Τρίτον, πολλοί συνάδελφοι μίλησαν για διαγραφή του σημείου 8. Να σας υπενθυμίσω πως ε, μεταξύ 72 και 80% των εμπορευματικών μεταφορών γίνονται στους δρόμους και όμως δεν υπάρχει μια υπηρεσία για αυτή την υπόθεση. Δεν πρέπει να το παραμερίσουμε τόσο εύκολα. Αλλά και εγώ δεν θα ήθελα τώρα να υπάρξει μια τέτοια υπηρεσία. Ως 100, ε, στην τροπολογία 105 έχω προτείνει μια μέση οδό. αναφέρθηκαν κάποιες υφτάμενες υπηρεσίες, ε, το Eurocontrol Route ε, και άλλες ε, για να βοηθήσουν στην εφαρμογή των νόμων. Οι αρχές αυτές τροχέας θα βοηθήσουν σε ευρωπαϊκή έναρμόνιση καθώς σήμερα υπάρχουν κάποιες ασάφειες και είναι τελείως διαφορετική ερμηνεία της υφιστάμενης νομοθεσίας. Οπότε εγώ θεωρώ πως πρέπει να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη στην τυποποίηση της ε, τεχνικής γνώσης, τη συγκέντρωση δεδομένων, τις πλατφόρμες ε, για τα δεδομένα αυτά. Η υποστήριξη αυτή υπάρχει ήδη σήμερα μέσω της ε, Eurocontrol Route και της Discol, αλλά δεν συμμετέχουν εκεί όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε, εγώ θα χαιρόμουν εάν ε, η ενισχυμένη συνεργασία την οποία πρότεινα στην 195 την τροπολογία μέσω της TISPOL και της Eurocontrol Route ε, εφαρμοστεί. Ευχαριστώ. τα πάντα. Έχω κατάλογο ολόκληρο και ε, αυτό το κατάλογο ακολουθώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θέλω και εγώ να ρίξω λάδι στη φωτιά. Σήκωσα το χέρι μου την ίδια στιγμή με άλλους συναδέλφους, αλλά άλλοι συνάδελφοι που είχαν σηκώσει την ίδια στιγμή με μένα το χέρι, μίλησαν εδώ και πολλή ώρα. Τέλος πάντων. Το βασικό είναι ότι μπορώ να μιλήσω. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για τη θαυμάσια δουλειά που έκανε, για όλη την προσπάθεια που έκανε για να εναρμονίσει τις προτάσεις όλων των συναδέλφων, ανεξάρτητα από την πολιτική του ομάδα. Είναι πολύ περιπλοκή η συζήτηση αυτή αλλά είναι και μια περίπλοκη πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Είναι αναγκαίο να ορίσουμε καλύτερα τον όρο αυτό κοινωνικό ντάμπινγκ. Δεν ξέρω αν είναι πρόθεση του εισηγητή να το κάνει σε αυτή την γνωμοδότηση, αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να μας παρουσιάσει ένα σαφέστατο ορισμό για το τι είναι το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρώπη διαπίστωσα ότι η συζήτηση για το κοινωνικό dumping έγινε μια συζήτηση για το κατά πόσον πρέπει να φτιάξουμε μια ευρωπαϊκή εταιρεία για τις οδικές μεταφορές. Ο κ. Κόρας πριν από μένα είπε ότι το 80% των ευρωπαϊκών μεταφορών γίνονται στο δρόμο. Χερσαίος και οι χερσαίες μεταφορές είναι ο μοναδικός τρόπος μεταφορών που δεν έχει αυτή τη στιγμή δική του υπηρεσία που θα ρυθμίζει τις δραστηριότητες του. Νομίζω ότι χρειάζεται μια τέτοια υπηρεσία και δεν πρέπει να καλυφθεί από ας πούμε μια υπηρεσία για τους σιδηροδρόμους ή για τις εναέριες μεταφορές ή για τις θαλάσσιες μεταφορές. Όχι, πρέπει να έχουμε μια δική μας υπηρεσία για τις χερσαίες μεταφορές πρέπει να εξηγήσουμε γιατί υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο. Γιατί είναι σύνθετες οι χερσαίες μεταφορές είναι και είναι σημαντικές. Γιατί έχει σημασία για την υγεία των εργαζομένων. Έχει σημασία γιατί μια τέτοια υπηρεσία θα βοηθήσει για να υπάρξει εναρμόνιση των κανόνων στην Ευρώπη και να θα φροντίσει για την εφαρμογή τους η υπηρεσία αυτή θα μπορέσει μέσω των δραστηριοτήτων της να βοηθήσει στην εναρμόνιση λοιπόν της νομοθεσίας. Και με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύονται καλύτερα οι οδηγοί και κυρίως οι επαγγελματίες οδηγοί. Αυτή τη στιγμή κάθε χώρα καθορίζει τους ελάχιστους μισθούς μόνη της και Αυτοί οι μισθοί αφορούν είτε τους ντόπιου εργαζόμενους ή τους ξένους που δουλεύουν στη συγκεκριμένη χώρα. Αλλά μπορούν κάποιες εταιρείε να προσλάβουν ε, οδηγούς, κυρίως ε, οδηγού από τις χώρες Ανατολική Ευρώπη και να τους αναγκάσουν να δεχτούν συμβάσεις και μισθούς με βάση το τι ισχύει στη χώρα πρόέλευσή τους. Θα πρέπει να μπει τέρμα σε τέτοιε πρακτικέ. Εάν πούμε όχι ότι υπάρχουν διαφορές ε, μισθών μεταξύ χωρών, αλλά, ανεξάρτητα από το ποια είναι η χώρα θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο κατόφλι κάτω από το οποίο δεν πρέπει να πέσουμε και αυτό το κατόφλι θα αφορά και τους ντόπιου εργαζόμενους και τους ξένους που δουλεύουν στη συγκεκριμένη χώρα. Επίσης, το βασικό είναι πώς θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τις πρακτικές ε, δυτικών εταιριών που προσλαμβάνουν εργαζόμενους, παραδείγματο χάρη οδηγού από την, ε, τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης με συμβάσεις και μισθούς αντίστοιχους με αυτούς που υπάρχουν στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Πρέπει να δει τέρμα σε κάτι τέτοιο. Όποια και αν είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μπει τέλος αυτή την πρακτική. Θα πρέπει να, βρει, να βρεθεί μια λύση, θα πρέπει να υπάρχει μια αρχή που θα εξασφαλίζει μια μεγαλύτερη εναρμόνιση της νομοθεσία και καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας. Τζος, όχι Γκεζίνε πάλι. Εντάξει, θα, δεν θα περιμένεις πολύ ώρα, Τζορτς, θα μιλήσω σχετικά σύντομα. Νομίζω ότι πολλές από τις συμβασικές τροπολογίες πήγαιναν προ τη σωστή κατεύθυνση για τα κοινωνικά θέματα. Δεν είμαστε ποτέ ομόφωνοι βέβαια, αλλά είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι έχουν σωστές συνθήκες εργασίας και οι εργαζόμενοι. Αλλά δεν μπορούμε να καταφερόμαστε και πάντα κατά των εργαζο... Ε, εργοδοτών, γιατί χωρίς τους εργοδοτές δεν μπορούμε ποτέ να καταλήξουμε σε μια πραγματικά εξισορροπημένη προσέγγιση. Εγώ θέλω να επενέσω την συμβαστική τροπολογία. 16 φυσικά περιλαμβάνει και τη δική μου τροπολογία. Δεν είναι, είναι τυχαίο και αυτό ίσως. Και είναι σημαντικό γιατί προηγουμένως το κείμενο είχε ένα κάπως ε, προστατευτικό χαρακτήρα και αναφερόταν, καταφερόταν και κατά της TTIP και του κινδύνου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τόνισε το, την ανάγκη να, τόνισε το, την ανάγκη να υπάρχουν ευρωπαϊκά πληρώματα στα πλοία και να φέρουν την ε, ε, ευρωπαϊκή σημαία, αλλά τώρα νομίζω τα πράγματα όπως την έχουμε αναδιατυπώσει τη 16 είναι πολύ καλύτερα. Ο Τζος Μπαχ έχει το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να χαιρετήσω το γεγονός ότι έχουμε επαρκή χρόνο να συζητήσουμε αυτή την γνωμοδότηση, δεν γίνεται πάντα κάτι τέτοιο. Αυτό είναι θετικό λοιπόν. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα φιλόδοξοι και θαραλέοι σε αυτήν την ε, γνωμοδότηση. Αναμένοντας το πακέτο για τις οδικές μεταφορές, και εδώ πρέπει να δώσουμε σαφείς κατευθύνσεις προς την Κομισιόν, που ελπίζουμε θα μπορέσει να τη συμπεριλάβει στο οδικό πακέτο. Γι' αυτό εγώ χαιρετίζω ιδιαίτερα το έργο του εισηγητή που έχει δημιουργήσει μια καλή γνωμοδότηση και επίσης και για τις ε, συμβαστικές τροπολογίες τις εκτιμώ ιδιαίτερα πηγαίνουν προς την καλή κατεύθυνση, σωστή κατεύθυνση. Δύο σημεία τώρα που θέλω να επισημάνω. Πρώτα απ' όλο, η σύνδεση των συνδικών εργασίας με την ασφάλεια. Έκανε σαφές εδώ ο εισηγητής ότι υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ των δύο και αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν αναγνωρίζεται πάντα ότι η ασφάλεια εξαρτάται και από τις σωστές εργασιακές συνθήκες. Πρέπει να τονίσουμε ότι το στρες, η υπερβολική κόπωση, όλα αυτά οδηγούν σε κινδύνους ατυχημάτων στους δρόμους, αλλά και σε άλλες μορφές μεταφορών, όπως έχουμε δει. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι το θέμα των ελέγχων. Και έρχομαι σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τελίτσα και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον ότι το πρόβλημα της ε, κατανομής αρμοδιοτήτων με τα κράτη-μέλη και της επικουρικότητος είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Δεν θέλω να θίξω την επικουρικότητα, αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο εν γνώση των προβλημάτων που προέρχονται από την ε, ποικιλομορφία στην εφαρμογή της νομοθεσίας και αυτό ιδίως σε χώρες όπου είναι πάρα πολύ σημαντικές οι διαμεθοριακές μεταφορές το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις και τρόποι εφαρμογής και εδώ πρέπει να, προσ... να εργαστούμε περισσότερο και επίσης το θέμα των ελέγχων. Η Κομισιόν έχει πει ότι θα εξασφαλίσει ένα ποσοστό ελέγχων, ένα ποσοστό αλλά αυτό δεν τηρείται από κανένα κράτος μέλος. Και κάποια κράτη-μέλη ουσιαστικά δεν δίνουν καθόλου ελεγκτικά δεδομένα. Δεν έχει στοιχεία για όλα αυτά η Κομισιόν. Επομένω, νομίζω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια να ασκήσει στα κράτη-μέλη πίεση ώστε να τηρούν την υποχρέωση να ασκούν αυτού του ελέγχου και συμφωνώ με αυτά που είπε ο Διδεκόχ. Βεβαίω πρέπει να υπάρχουν όχι μόνο έλεγχοι, αλλά να υπάρξουν και ουσιαστικέ κυρώσεις και όχι κάτι το οποίο μπορούν να το πληρώσουμε διότι είναι ασήμαντος ε, χρηματικό πρόστιμο. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στους ελέγχους και να βρούμε έναν τρόπο να βελτιώσουμε την κατάσταση, η οποία αυτή τη στιγμή έχει πολύ διαφορετική εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Ο κύριος Γουίλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του που έχει κρατήσει τις τελευταίες εβδομάδες αλλά και τους τελευταίους μήνες. Είχαμε πολύ έντονες συζητήσεις, πολλές φορές υπήρξαν πολλές τροπολογίες οι οποίες κατετέθησαν. Φυσικά κάποτε πρέπει να καλυφθούν από συμβαστικές τροπολογίες. Εγώ έχω υποβάλει νέα τροπολογίες και αυτές τις έχει συμπεριλάβει στις συμβαστικές τροπολογίες ο εισηγητής και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Ξέρω ότι είμαστε η Επιτροπή Μεταφορών και απλώς γνωμοδοτούμε προς την Επιτροπή Απασχόλησης. Αλλά νομίζω ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να εξηγήσουμε τι σημαίνει για μας το κοινωνικό ντάμπινγκ για την Επιτροπή Μεταφορών και για τον τομέα αρμοδιοτήτων μας. Το φαινόμενο αυτό δεν το αντιλαμβάνομαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο στις πολιτικές συζητήσεις που κάνουμε. Αυτό είναι ανάγλυφο. Στα διάφορα κράτη-μέλη υπάρχει μια διαφορετική χρήση αυτής της ε, έννοιας του κοινωνικού ντάμπινγκ. Όσο λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να έχουμε μια ενιαία αντίληψη, ένα ενιαίο ορισμό του κοινωνικού ντάμπιν, είναι πολύ δύσκολο εμείς να μπορέσουμε να εστιάσουμε αποκλειστικά και μόνο στον τομέα των μεταφορών που είναι η δική μας σφαίρα αρμοδιοτήτων. Γι' αυτό στις τροπολογίες μου, στην 42 παραδείγματος χάρη, έχω τονίσει αυτό το πρόβλημα, έχω τονίσει ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Επίσης στην τροπολογία 112 εγώ έχω αντιμετωπίσει ένα περαιτέρω πρόβλημα που και αυτό το έχουν θίξει άλλοι συνάδελφοι. Πρόκειται Πρόκειται για Πρόκειται για τα οχήματα τα οποία έχουν βάρος ωφέλιμο κάτω των 3,5 τόνων και εδώ τίθεται το θέμα των συνθηκών εργασίας των οδηγών τους. Για τους οδηγούς οχημάτων άνω των 3,5 τόνων υπάρχουν κανόνες οι οποίοι ισχύουν και εφαρμόζονται, είναι υποχρεωμένοι να έχουν κάποιες προδιαγραφές αλλά αυτές οι προδιαγραφές δεν έχουν εφαρμοστεί για τα μικρότερα οχήματα και δεν εφαρμόζονται. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται και για τα μικρότερα φορτηγά. Θα σήμαινε βέβαια και μεγαλύτερο γραφειοκρατικό βάρος, αλλά για μένα είναι μια πολύ καλή ιδέα. Σε ό,τι αφορά επίσης την συζήτηση που έχει λάβει η χώρα μέχρι στιγμής για τα θέματα αυτά, Η συζήτηση αυτή δεν οδήγησε, πιστεύω, σε μεγάλες αντιπαραθέσεις. Υπήρξαν πιο έντονες συζητήσεις ε, στο παρελθόν για τα θέματα αυτά. Για μένα το πρόβλημα πρέπει να το δούμε καταρχήν από την οπτική γωνία των εργαζομένων. Εγώ φυσικά είμαι σοσιαλιστής, ανήκω στην ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Θα ήθελα όμως περαιτέρω να πω ότι πιστεύω ότι οι συνάδελφοι από τη Δυτική Ευρώπη, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, πολλές φορές ενδιαφέρονται να προστατεύσουν τις ε, δικές τους εταιρείε την ε, δική τους αγορά και μόνο. Και να σας πω αυτό το παράδειγμα. Ένας Γάλλος ο οποίος προσπαθεί να προστατεύσει τη δική του αγορά προσπαθεί να εκδιώξει μέσα σε εισαγωγικά τις ε, κεντροανατολικές ε, εταιρείε από τον τομέα αυτό και φυσικά ο στόχος του είναι να εργάζονται οι οδηγοί από την κεντροανατολική Ευρώπη με, αποδοχή, με τις δικές τους αποδοχές στις δυτικές εταιρείε. Αλλά όταν γίνεται κάτι τέτοιο να τους πληρώνουν και λιγότερο από ό,τι θα πληρώνανε δυτικοευρωπαϊκούς εργαζόμενους. Εάν λοιπόν γίνεται κάτι τέτοιο, αν θέλουν μια babysitter παραγωγή χάρη για το σπίτι τους, προτιμούν μια κεντροανατολικό Ευρωπαία από μια Γαλλίδα γιατί θα τους κοστίσει φυσικά φθηνότερο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί υπάρχει και σύγκρουση ενδεχόμενη συμφερόντων που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Βιμ Φαντενκάμπ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το οποίο συζητάμε είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα του τομέα των μεταφορών. Ωραία είναι να μιλάμε για το ΣΕΦ και το ΕΦΣΙ και τους διαδρόμους διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, αλλά οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί πέρα έχουν μεγάλο πρόβλημα και πολλοί από εμά στην προεκλογική εκστρατεία του 2014 κατεβήκαμε με σύνθημα μια πιο κοινωνική Ευρώπη. Για πολλούς ανθρώπους η Ευρώπη είναι μια γραφειοκρατία τις Βρυξέλλες ε, που έχει ελάχιστη καμία σχέση με κοινωνικές πτυχές. Αυτό θεωρώ πως είναι καλό να το σκεφτούμε αυτό σήμερα. Η δεύτερη μου παρατήρηση, και εδώ επαναλαμβάνω λίγο αυτά τα οποία είπε ο Πολωνός συνάλφος, οι διαφορές των τιμών στην εσωτερική αγορά δεν είναι κοινωνικό dumping. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί η εσωτερική αγορά έχει διαφορές ποιότητας και τιμών. Και αυτό είναι ο πυρήνας της εσωτερικής αγοράς, δεν είναι κοινωνικό ντάμπινγκ. Θα το λέω συνέχεια αυτό. Αλλιώ θα γίνει χαμός αν το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Μετά έχουμε το εσωτερικό κοινωνικό ντάμπινγκ. Εντός του ΕΛΚ προφανώς ε, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ με αυτό το θέμα και οδηγούμαστε σε μια αυτοθυματοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δει κανείς Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, Νότια Αφρική, εμείς στην Ευρώπη με το μοντέλο του Ρήνου, όπως λέμε, Έχουμε ένα πολύ επιτυχημένο μοντέλο. Αυτό το οποίο λοιπόν πρέπει να προσέξουμε είναι να μην λέμε από μόνοι μας ότι είμαστε μπανανία, ότι δεν υπάρχει κοινωνική προστασία. Από τους 100 εργαζόμενους στις μεταφορές, 80% έχουν καλό εισόδημα, καλές κοινωνικές παροχές. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν όταν γράφουμε αντικοινωνικό dumping εδώ πέρα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα στον τομέα των μεταφορών. Απλούστατα δεν είναι αλήθεια. Ο κύριος Νίλσεν πρέπει να διακρίνει στην έκθεσή του αυτά τα δύο πράγματα. Τέλος, ο άλλος ε, όρος που ανέφεραν οι συνάδελφοι, ο κύριος Μπαχ και οι Λυπή. Η εφαρμογή. Έχουμε νομοθεσία δεν εφαρμόζεται. Τα κράτη-μέλη λένε ότι ναι θα τα κάνουμε και τα λοιπά, αλλά μετά στις χώρες δεν εφαρμόζεται. Έχετε επαφές με το ETF, ε την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις και μας λένε δεν θέμε νέα νομοθεσία, θέμε εφαρμογή της υφιστάμενης. Και τέλος, για το European Road Agency θα συμφωνήσω με τον κύριο Φαντάλεν. Τι μπορεί να σημάνει εδώ πέρα το Eurocontrol. Κανείς δεν θέλει άλλη μία γραφειοκρατία. Και μην ξεχνάτε πως η εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας εξακολουθεί ακόμα να είναι στην επικουρικότητα, δεν έχει αρμοδιότητα η Ένωση. Είναι ζήτημα επικουρικότητας, να υπάρχει ευρωπαϊκή συνεργασία, εδώ πέρα μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο το Eurocontrol για τους δρόμους. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ισμαήλ Ερτούγ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά ακούστηκαν. Ο Γιάννης Νίλσεν νομίζω εδώ πέρα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και εξακολουθεί να το κάνει και πρέπει να το κάνει γιατί θεωρώ ότι είδαμε στα τελευταία λεπτά πόσο διαφορετική είναι η εικόνα που υπάρχει εδώ στην αίθουσα για την κατάσταση όταν παραδείγματο χάρη λέμε ότι το Πέτερ Φαντάλεν λέει να μην το δούμε ιδεολογικά. Μα συμφωνώ απολύτω. Να μην το δούμε ιδεολογικά, να δούμε την πραγματικότητα σήμερα. Η πραγματικότητα είναι όταν λέμε πως υπάρχουν διαφορές τιμών στην εσωτερική αγορά και ότι αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ε, κοινωνικό ντάμπινγκ. τότε αντιλαμβάνομαι, εντάξει, μια κάποια λογική, αλλά μετά εμείς είμαστε αυτοί μετά που κατηγορούμε την Emirates ε, και την Etihad ότι έχουν χαμηλές τιμές για να μπουν στις αγορές μας. Αυτό είναι social dumping. Ότι όταν γίνεται όμως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι social dumping, κοινωνικό dumping εντάξει, να το δούμε λίγο σοβαρά. Νομίζω πρέπει να το δούμε κάπως αλλιώς. Και πράγματι συμφωνούν όλοι από δεξιά με χρειάζεται, ότι χρειάζεται ένας ορισμός. Να δούμε λοιπόν την κατάσταση και να αναφερθώ λίγο στους ε, συντηρητικούς φίλους, ότι αυτό, αυτοί οι ίσοι όροι ανταγωνισμού που επικαλούνται σημαίνουν πως θα πρέπει να υπάρχει σωστή νομοθεσία και στον τομέα αυτών. Και δεν ξέρω Βιμ ε, με ποιους ε, αρμόδιους μίλησε εσύ στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση Οδικών Μεταφορών, αλλά εκεί πέρα εγώ με αυτούς μίλησα μου είπαν ότι υπάρχει κοινωνικό ντάμπινγκ και θέλουν να βοηθήσουμε, ειδικά στην εφαρμογή. Και έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα εδώ στην Κομισιόν. Γιατί η Κομισιόν δεν τα εφαρμόζει. Είναι θεματοφύλακα των συνθήκων, έχει όλα τα μέσα. Και βλέποντας το τι κάνει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και το πόσο γρήγορα κινείται σε κάποιες ε, διαδικασίες, αναρωτιέμαι γιατί εδώ πέρα κάθεται επί χρόνια και κοιτάει. Είναι πολύ γνωστές οι χώρες που δεν εφαρμόζουν κάποια πράγματα που έχουν συνυπογράψει. Και ε, πραγματικά αναρωτιέμαι και μετά αναρωτιόμαστε γιατί στις εκλογές ε, κάποιοι ψηφοφόροι πάνε στους ε, ρατσιστές. Δεν ναι, γιατί τα λένε αυτά όμως. Για τα δικά τους κίνητρα, αλλά τα φύγουν. Και όταν θέλουν να διαμαρτυρηθούν οι ψηφοφόροι, αυτό κάνουν. Οπότε δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικής διάστασης ή ιδεολογίας, όχι είναι νομίζω το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα κάνουμε με την ευημερία των πολιτών, των εργαζομένων κυρίως. Πριν από 1,5 χρόνο, μετά τις ευρωεκλογές, όταν βγήκε ο κύριος Γιούνκερ και μας είπε ξεκάθαρα, πιο καθαρά από οποιονδήποτε άλλον πρόεδρο της Κομισιόν, ότι πρέπει να δούμε την κοινωνική Ευρώπη. Θεωρώ πως ε, ίσως ε, δεν τον κατάλαβαν τα κόμματα, ε, τα δικά του έτσι, τα συντηρητικά, οι δικές του κυβερνήσεις. Γι' αυτό θα ήθελα να απευθυνώ μια έκκληση πραγματικά στον τομέα του, των ίσων όρων ανταγωνισμού που λέτε, να φροντίσουμε να στηρίξουμε και τις επιχειρήσεις μας και να μην τιμωρήσουμε αυτούς οι οποίοι τηρούν τελικά τον νόμο, την ώρα οδήγησης και ανάπαυσης. Αυτοί οι οποίοι πληρώνουν σύμφωνα με τις συλλογικέ συμβάσεις και που δίνουν τις άδειε. Μην τους τιμωρούμε κιόλας. και να μην τα βλέπουμε αυτά ως ε, ιδεολογία, είναι realpolitik, ξεκάθαρα. Για να κλείσει κάπως αυτή η ψαλίδα. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Μην ξεχνάμε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία είναι ένας από τους πυλώνες βασικής ένωσης. Είναι σημαντικό και οικονομικά και πολιτικά κάτι τέτοιο. Είναι μία από τις μεγαλύτερες ε, ελευθερίες και τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυκλοφορία των εργαζομένων, των αγαθών και των κεφαλαίων. 280 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το κέρδος από την ελεύθερη κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ελευθερία. Αφορά την ε, ενιαία αγορά και χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερη κυκλοφορία. Περισσότερη ελευθερία στην κυκλοφορία των ανθρώπων και των αγαθών. Δεν πρέπει να δημιουργούμε περισσότερους φραγμούς. Στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκής Ένωση προφανώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μισθών. Είναι σημαντικό όμω να έχουμε σαφεί κανόνε για τι είδους ανταγωνισμό έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλίσουμε την οδική ασφάλεια. Γι' αυτό τα οχήματα να είναι, θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, να έχουν καλούς οδηγούς και να εξασφαλίσουμε καλές συνθήκες εργασίας. Θα πρέπει να έχουμε επαρκή νομοθεσία που εξασφαλίζει αυτές τις ε, συνθήκε εργασία. Νομίζω όμω ότι έχουμε του κανόνε. Έχουμε την νομοθεσία. Αρκετή νομοθεσία για την οδική ασφάλεια. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι έλεγχο των κανόνων. Δεν θέλουμε αντίθετα φράγματα στην κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών. Το επόμενο θέμα αφορά την υπηρεσία αυτή οδικών μεταφορών. Είμαι πολύ επικριτική για κάτι τέτοιο. Δεν θέλω να αντιμετωπίζουμε έτσι τα προβλήματα, να δημιουργούμε νέου οργανισμού, νέε υπηρεσίε. Όταν έχουμε προβλήματα, δεν νομίζω ότι τα λύνουμε με μια νέα υπηρεσία. Ειδικά στον τομέα των μεταφορών, δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε τομεακέ υπηρεσίε. Θα πρέπει να θεωρούμε ότι οι μεταφορέ είναι ένα όλο. Οι θαλάσσιες, οι εναέριε, οι χερσαίε και οι συρδομικέ. Είναι ένα όλο, ένα πακέτο. Δεν χρειαζόμαστε υπηρεσίες ανά συγκεκριμένο τρόπο μεταφορών. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η προηγούμενη συνάδελφος για την ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Ντεμόντε. Έχει νόημα αυτή η εσωτερική αγορά, γιατί δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τον ανταγωνισμό. Είναι σαφές όμως ότι ο ανταγωνισμός θα πρέπει να βασίζεται σε παραγωγικές συνθήκες που είναι παρόμοιες. Αυτό απαιτεί φυσικά χρόνο. Αν δεν καταφέρουμε όμως να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο, τότε φιλολογούμε απλώς, μένουμε στη θεωρία και δεν περνάμε στην πράξη. Και επομένως η ευρωπαϊκή οικοδόμηση θα μείνει μετέωρη. Σε ό,τι αφορά τις οδικές μεταφορές, έχουμε κάποιες χώρες όπου οι εταιρείε ε, οδικών μεταφορών έχουν, αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος λόγω ε, της τιμής των καυσίμων και άλλοι αντιμετωπίζουν ψηλότερο κόστο λόγω της, ε, ε, των μισθών, δηλαδή το πόσο καθίσει το, τα εργατικά. Και παίζουμε γύρω από αυτά. Τι κάνουν λοιπόν οι εταιρείε οδικών μεταφορών. Προσπαθούν να μειώσουν τις τιμές, αλλά όπως είπαν και διάφοροι συνάδελφοι, προσπαθούν να αυξήσουν το χρόνο εργασίας των εργαζομένων τους, ε, παρακάμπτοντας τους κανόνες ε, για την ανάπαυση τα λοιπά και πέσοντας με τους ε, ταχυγράφους. Αυτό συμβαίνει και στην, ε, στις μεταφορέ, μεταφορές. Το ακούσαμε και στην ακρόαση. Ακούσαμε ότι υπάρχουν πρακτικές όπου η, αυτόνομη, η ψευδής αυτόνομη εργασία ε, χρησιμοποιείται και βεβαίω έχει αρνητικέ επιπτώσει για την ασφάλεια. Τι μπορούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε φυσικά αυτέ τι πρακτικέ, να βρούμε νέου τρόπου ε, ε καταγραφή του χρόνου εργασία, νέου ταχυγράφου. Και βεβαίω να παίξουμε πάνω στους, ε, και να δούμε πώ μπορούμε να βελτιώσουμε του ελέγχου. Συγχαίρω μάλιστα τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητέ για τη δουλειά που κάναν προς αυτή την κατεύθυνση και για τον υψηλό αριθμό συμβαστικών τροπολογιών για να υπάρξει συμφωνία. Αλλά σήμερα οι εθνικοί έλεγχοι αφορούν τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των εθνικών ε, επιχειρήσεων. Υπάρχει πρόβλημα. Τι γίνεται με τις υπόλοιπες. Γι' αυτό έχουμε πολλά να κάνουμε, πολλά να κάνουμε ακόμα. Επίσης, οι κυρώσεις ή θα είναι αποτρεπτικές ή δεν έχουν κανένα νόημα όπως οποιοδήποτε νομικό μέτρο. Ε, εάν δεν είμαστε σε θέση να το πετύχουμε αυτό, να έχουμε αποτελεσματικούς ελέγχους, θα πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση σε σχέση με το καμποτάζ, να μειώσουμε τις εθνικές μεταφορές ή να υπάρχουν εμπρό πίσω ας πούμε ε, ή να εξασφαλίσουμε την απόσπαση των εργαζομένων. Θα πρέπει να έχουμε μια πολύ ρεαλιστική προσέγγιση γιατί εκεί παίζεται η παραγωγικότητα και δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτό το πρόβλημα και να μην βρούμε λύση. Ευχαριστώ. Και εγώ ζήτησα να λάβω το λόγο τώρα. Είναι σημαντικά τα κοινωνικά θέματα, προφανώς. Και έχει γίνει σαφές τώρα από τις τελευταίες στατιστικές ότι 36 άνθρωποι έχουν την ίδια περιουσία που έχει το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού περίπου, 36 οικογένειες. Είναι όλο και περισσότεροι οι πλούσιοι και είναι όλο και περισσότεροι οι φτωχοί. Υπάρχουν αρκετά χρήματα μεν, αλλά το θέμα της διανομής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προφανώς εδώ πρέπει να υπάρχει η αρχή της ίσης αμοιβή για ίση εργασία. Αυτό είναι στοιχείο της νομοθεσίας. Αλλά υπάρχουν εδώ διαφορές μεταξύ των κρατών της Ευρώπης. Όταν βλέπουμε παραγωγής χάρη ένα μιας ε, ε νοσοκόμα στη Σουηδία που πηγαίνει στην Νορβηγία για να βγάλει περισσότερα λεφτά αλλά εργάζεται με τις συνθήκες που δουλεύουν και οι νοσοκόμες στην Σουηδία, αυτό είναι εντάξει. Αλλά αν δούμε τώρα τις περιπτώσεις των Πολωνών, ε, Ραβλικών και της ε, αντίδρασης που έγινε, που δημιουργήθηκε τότε. Μα χρειάζονται αυτοί να δουλεύουν και στην Πολωνία και να βρίσκονται και εκεί οι αποδοχές τους στο ίδιο επίπεδο. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντική η αρχή της ίσης αμοιβή για ίση εργασία. Και εδώ φυσικά είναι απαραίτητο όταν υπάρχουν παραβιάσεις να υπάρχουν και κυρώσεις. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ να πάω σε ένα νοσοκομείο στο Μόναχο ή στο Βερολίνο που η, Βουλγα, η Βουλγάρα νοσοκόμα πληρώνεται λιγότερο από την Γερμανίδα συνάδελφό τη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεικτο. Αλλά ακόμα και μέσα στι χώρε υπάρχουν διαφορέ. Εγώ έρχομαι από το Βερολίνο. Και στο Βερολίνο παίρνουν λιγότερα λεφτά οι δάσκαλοι, παραδείγματο χάρη, οι καθηγητέ, 100 ευρώ λιγότερα από ότι από αυτού που βρίσκονται στο Βραδεμβούργο. Αυτό είναι θέμα βλακείας ή θέμα ευφυΐας ίσως για ορισμένους, αλλά είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν τα ίδια δικαιώματα και οι ίδιες αμοιβέ για όλους. Αυτά που είπατε λοιπόν είναι απαραίτητο να γίνουν πραγματικότητα και πιο έντονη έλεγχη και να υπάρχουν και κυρώσεις. Έχουμε αγωνιστεί για το χρόνο ανάπαυσης των οδηγών των φορτηγών να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο και μία εφαρμογή και αστυνόμευση. Λοιπόν, περιμένουμε από την Κομισιό να κάνει κάτι για να τα ελέγξει όλα αυτά. Εσείς είστε ο θεματοφύλακας των συνθήκων. Δεν μπορείτε να αφήνετε να παραβιάζονται οι συνθήκες και να αφήνετε τους δράστες να μην κάνουν τίποτα. Αμα είναι έτσι δεν έχει κανένα νόημα να νομοθετούμε αν ακόμα και τους νόμους που έχουμε περάσει εσείς δεν θέλετε να τους εφαρμόσετε και ούτε υπάρχει καμία εγγύηση με τη δημιουργία νέων φορέων ή νέας νομοθεσίας <clears throat> να εξασφαλίσουμε την ε, εφαρμογή. Για τις ε, πρακτικές λύσεις. Αναφέρθηκε η συζήτηση που κάναμε με τους οδηγούς των φορτηγών. Υπάρχει αυτή η περίπτωση του οδηγού από την Ρωμανία, ο οποίος 8 μήνες δεν πάτησε το πόδι στη Ρουμανία. Γύρισε μονάχα σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης και έπαιρνε τον ελάχιστο μισθό της Ρουμανίας 250 ευρώ και πληρωνόταν με το χιλιόμετρο, όχι με τις ώρες που δούλευε. Δηλαδή αν έμενε μια ώρα σε μποτιλιάσμα ήταν δικό του πρόβλημα, δεν έπαιρνε πεντάρα γιατί πληρωνόταν μονάχα με το χιλιόμετρο. Αυτό είναι απόλυτα παράδεκτο. Και εδώ υπάρχουν πρακτικές λύσεις. Υπήρξε, όπως είπε η εκπρόσωπος της ε, Ένωσης των Εργατικών Ενώσεων να υπάρχει εφαρμογή ταχογράφων. Αυτό επιτρέπει την εφαρμογή της ομοθεσίας. Και αυτό έχει γίνει δεκτό από την Κομισιόν με τη λεπτομέρεια ότι μόνο σε 20 χρόνια θα είναι πλήρης η εφαρμογή. Λοιπόν, οι πρακτικέ λύσει υπάρχουν, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε 20 χρόνια για να τις εφαρμόσουμε, γιατί μέχρι τότε θα έχουν καταστραφεί όλα αυτά τα οποία δημιουργήσαμε τα τελευταία 50-60 χρόνια στην Ευρώπη. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι όλε αυτέ οι πρακτικέ λύσει οι οποίε υπάρχουν σήμερα να εφαρμοστούν ώστε να σταματήσει αυτό το κοινωνικό dumping. Δεν είναι όλοι βέβαια απαταιώνε, αλλά θα πρέπει αυτοί οι οποίοι καταχρώνται και παραβιάζουν τους κανόνες να είναι σε, είμαστε σε θέση να τους να επιβάλλουμε κυρώσεις. Πρέπει να ασκηθεί λοιπόν η αρχή ότι ίση αμοιβή για ίση εργασία και θα πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες κυρώσεις για να αποτρέψουν αυτούς που θέλουν να ε, παραβιάζουν τους κανόνες. Και τέλος δίνω το λόγο τώρα στην Κομισιόν. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Δύο γενικέ παρατηρήσει για το σχέδιο έκθεση και για τι συμβαστικέ τροπολογίε του εισηγητή. Και θα ήθελα επ' να αναφέρω πολύ σύντομα κάποια σημεία για κάποιε από τι συμβαστικέ τροπολογίες. Να ξεκαθαρίσω ότι εκφράζω προκαταρτικές απόψεις Κομισιόν και η επίσημη άποψη της Κομισιόν για το σχέδιο έκθεσης και για τις τροπολογίες δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί. Ας ξεκινήσουμε με τις δύο γενικές παρατηρήσεις. Πρώτον, ελπίζω έτσι να απαντήσω και την ερώτηση που μας απευθύνεται για την έννοια του κοινωνικού τάμπινγκ, που είναι και το αντικείμενο του Συμβασμού Υπαριθμών 6 της, του εισηγητή. Η Κομισιόν πιστεύει ότι είναι δύσκολο και επίμαχο το θέμα αυτό, είναι δύσκολο να το ορίσουμε. Δεν θέλω να πω ούτε καν ότι θα ήταν και επικίνδυνο να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε με νομικές υποχρεώσεις και με κυρώσεις την τήρηση κάποιων αρχών γύρω από την ακύρωση του κοινωνικού ντάμπινγκ. Ο κ. Ζήλερ και διάφοροι άλλοι μίλησαν για την τροπολογία 17. Λέει ότι δεν υπάρχει σαφής και καθολικά αποδεκτή άποψη για το κοινωνικό ντάμπι και ερμηνεύεται διαφορετικά αυτός ο όρος και αυτό μπορεί να δημιουργήσει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει το υπόλοιπο, μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση και μερικές φορές να ενσωματώσει και να συμπεριλάβει και προστατευτικά μέτρα που μπορεί να οδηγήσει στην κατακαιρμάτιση της ενιαίας αγοράς. Αυτό είναι η άποψη και της Κομισιόν. Η Κομισιόν δεν αρνείται βεβαίως ότι το φαινόμενο του κοινωνικού ντάμπινγκ υπάρχει και καλό θα ήταν, ένα άλλο θέμα είναι το να προσπαθήσουμε νομικά να το προσδιορίσουμε. Αλλά το πιο σημαντικό για την Κομισιόν είναι το εξή. Είναι μάλιστα διτή, διτό το θέμα. Πρώτον, ε, σαφείς κανόνες για την πρόσβαση στο επάγγελμα, για πρόσβαση στην αγορά, ε, για το χρόνο εργασία, σαφή κριτήρια για να... Σαφείς κανόνες για για τις εταιρείε μεταφορών και στον τομέα των οδικών μεταφορών και στον τομέα της των εναέριων, της κυκλοφορίας και θα πρέπει να επιβάλλονται κανόνες αυτοί και με αποτρεφτικά μέτρα, δηλαδή κυρώσεις, ε, κανόνες και καλή πολιτική εφαρμογής. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον καλύτερο τρόπο το κοινωνικό ντάμπινγκ, χωρίς την ανάγκη να προσπαθούμε να επινοήσουμε ένα νέο ορισμό για αυτή την έννοια. Για το συμβασμό 6 να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαστε υπέρ της δημιουργίας αυτού του μαυροπίνακα ε, των ε, εταιριών οδικών μεταφορών. Δεν είμαστε υπέρ αυτού του εργαλείου που μοιάζει ωραίο, αλλά δεν θεωρούμε ότι είναι κατάλληλο εργαλείο για να βελτιώσουμε την ε, εφαρμογή των κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερη γενική παρατήρηση για την έκθεση αυτή. Το ξανασυζητήσαμε μάλιστα σε προηγούμενες συνεδριάσεις. Είναι η ανάγκη να έχουμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα σε διαφορετικούς ε, στόχους της συνθήκης. Απ' τη μία θα πρέπει να προωθήσουμε την εσωτερική αγορά και την αρχή της ε, ελευθερίας παροχής υπηρεσιών και από την άλλη την αρχή της κοινωνικής προστασίας και του δίκαιου ανταγωνισμού. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα σε αυτούς τους στόχους. Ο συμβιβασμό υπαρχών 2 του εισηγητή κινείται προς αυτή την κατεύθυνση ακριβώς. Σύντομα θα ήθελα να αναφέρω τώρα κάποιες από τις συμβαστικές τροπολογίες. Η νούμερο 7 που ζητάει από την Κομισιόν και από τα κράτη-μέλη να περιορίσουν τις διαφορές μορφές άτυπης απασχόλησης που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια. Θα ήθελα να αναφέρω σε αυτό ότι η Κομισιόν υιοθέτησε στις 8 Μαρτίου μια πρόταση για να θεωρήσει την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων και παράλληλα έχει ξεκινήσει μια δημόσια διαβούλευση για το, τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Κεφάλαιο 2 αυτής της διαβούλευσης για τις ε, δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού που, μιλάει, που μιλάει για τη νέα μορφή απασχόλησης, την ευέλικτη απασχόληση ε, γι' αυτή θα πρέπει να ενημερώνονται καταλήλως οι εργαζόμενοι και οι εργοδότε είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν αυτή την ενημέρωση. Συμβασμό 9 που αφορά την ανάγκη Κομισιόν να ετοιμάσει ένα ηλεκτρονικό αρχείο για όλους τους, ε, τις εταιρείε που λειτουργούν με κοινοτική άδεια. Προσοχή, πριν επινοήσουμε νέα εργαλεία, γιατί ήδη έχουμε πολλά που υπάρχουν και θα πρέπει απλώς να τα εκμεταλλευτούμε. Σας παραπέμπω στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ε, Ευρωπαϊκό Συγγνώμη Μητρό, απατών ε, από εταιρείε μεταφορών. Πριν από μερικέ εβδομάδε ήρθα εδώ μπροστά σα για να σα παρουσιάσω ένα σχέδιο κανονισμού για να βελτιώσουμε την λειτουργία ακριβώς αυτού του Μητρώου και στο μέλλον το Μητρό αυτό θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών για τις άδειε των ε, εταιριών οδικών μεταφορών. Πριν δημιουργούμε λοιπόν νέα εργαλεία, σας παρακαλώ ας αξιολογήσουμε τις ανάγκες για αυτές τις για τη δημιουργία τέτοιων ε, εργαλείων. Επίσης, πολύ σύντομα να αναφέρω και τον συμβασμό 10 για την ανάγκη να αξιολογήσουμε τα κράτη-μέλη όπου χρησιμοποιούν πάρα πολύ ε, τις εταιρείες οδικών μεταφορών. Το αναφέρετε και εσείς, Πρόεδρε, αυτό το θέμα. Είναι κάτι το οποίο αξιολογούμε στα πλαίσια της αναθεώρησης της νομοθεσίας για τις οδικές μεταφορές. Η τροπολογία αφορά τις εταιρείες ε, γραμματοκιβώτια. Επίσης, ε, συμβασμός 14 για τον ε, κοινωνικό, το κοινωνικό dumping των εταιριών εναέρειας κυκλοφορίας. Δεν θέλω να το σχολιάσω λεπτομερώς, αλλά η νέα διατύπωση της νέας τροπολογίας, της τροπολογίας αυτής πηγαίνει προς την κατεύθυνση. Επίσης, συμβασμός 17 για το θέμα της μεταφοράς προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής ε, παρόχου, εταιρείας δηλαδή. Η τροπολογία αυτή είναι νέα. Η Κομισιόν δεν είναι υπέρ αυτής της τροπολογίας και αυτό το θέμα το συζητάμε και στα πλαίσια του τέταρτου συνδρομικού πακέτου δεν είναι υπέρ μιας ε, γενικής υποχρέωσης για τη μεταφορά προσωπικού. Αυτό το, το θέμα ρυθμίζεται στην οδηγία του 2001 κάθετο 23 και πιστεύουμε ότι ξεπερνάει τα όσα προβλέπει αυτή η οδηγία. Και αν ε, ξεπερνάμε την ε, οδηγία αυτή θα πρέπει να αποφασίζεται περιπτωσιολογικά σε εθνική βάση ή μέσω συλλογικών συμβάσεων. Δεν βλέπω ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτή τη τροπολογία σε σχέση με αυτά που υπάρχουν ήδη στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, στην Οδηγία δηλαδή. Και να τελειώσω την παρέμβασή μου απαντώντα σε δύο ερωτήσει που απευθύνθηκαν στην Κομισιόν. Πρώτον, για την Οδηγία Απόσπαση των Εργαζομένων. Η, η Κομισιόν υιοθέτησε μια πρόταση στι 8 Μαρτίου για τη νέα οδηγία και εκεί αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή αυτή τη οδηγία τι οδικές μεταφορές έχει δημιουργήσει πολλές ε, δυσκολίες και αναγγείλαμε ότι πρέπει να ανάγκη να διευκρινίσουμε την εφαρμογή της οδηγίας αυτής στις οδικές μεταφορές. Είμαστε σε φάση αξιολόγησης ακόμα. Πώς θα το κάνουμε, πώς θα την αξιολογήσουμε αυτή την οδηγία για τις οδικές μεταφορές, τι διευκρινήσεις θα κάνουμε, δεν είμαστε σε θέση σήμερα να σας πούμε περισσότερα αλλά είναι κάτι που δεν το ξεχνάμε. Τελευταίο σημείο. Το γενικό θέμα της εφαρμογής που ακούστηκε πολλές φορές, κυρίως για τον καονισμό του 2006-561 για την οδήγηση και ανάπαυση των επαγγελματιών οδηγών. Είμαστε σε φάση αξιολόγησης αυτού του καονισμού του 2006 δεν έχει τελειώσει η αξιολόγηση. Δύο πράγματα όμως έχουν προκύψει από, τα, από την αξιολόγηση που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Πρώτον, χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες. Και με βάση αυτά τα προκαταρτικά αποτελέσματα φαίνεται ότι κάποιοι κανόνες δεν είναι τόσο σαφείς όσο θα έπρεπε. Δεύτερον, που προκύπτει επίσης σαφώ από την αξιολόγηση, είναι η ανάγκη να βελτιώσουμε την εφαρμογή. Η πρώτη ευθύνη για την εφαρμογή βαραίνει τα κράτη-μέλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση νίτη τα σχήρα τη. Βεβαίω, μπορούμε να εξασφαλίσουμε την προσθέμενη αξία στην εφαρμογή, βελτιώνοντα την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών εφαρμογής και με τη βελτίωση του συντονισμού ανά, ανάμεσα στις αρχές αυτές. Αυτό είναι το αντικείμενο της πρωτοβουλίας που ετοιμάζουμε για τις οδικές μεταφορές. Επίσης, ερευνούμε πολλές υποθέσεις παραβιάσεων. Δεν μπορείτε να μας κατηγορήσετε ότι δεν κάνουμε τίποτα. Μπορούμε να βελτιώσουμε αυτά που κάνουμε αλλά να σας δώσω και κάποια παραδείγματα. Όποτε ακούμε παράπονα για εταιρείε ε, γραμματοκιβώτια, σας διαβεβαιώ παρότι δεν είναι γνωστό Εβραίος, ότι κάνουμε, ε, απευθύνουμε ένα αίτημα προς το κράτος μέλος για να διερευνήσει το θέμα και για να ελέγξει αν πραγματικά μια εταιρεία είναι εγκατεστημένη στο έδαφος του εν λόγω κράτου μέλους ή είναι απλώς εταιρεία γραμματοκιβώτιο. Ευχαριστώ, ο Μάρκος Πίπερ ζήτησε το λόγο. Κοιτάξτε τώρα. Έχω εκπλαγεί λίγο. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες μας εδώ στο πρόσωπο της Κομισιόν, αλλά Αυτές είναι μόνο συμβαστικές προτάσεις ε, του εισηγητή. Εμείς τι να καταλάβουμε από αυτά. Οπότε φαίνεται υπάρχει δηλαδή ήδη μια συμβαστική λύση η οποία είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση και η Κομισιόν τοποθετείται ήδη. Το αμφισβητώ αυτό. Και δεύτερον, να αρχιέμαι με τον τριμερή διάλογο. Είχαμε την εντύπωση πως η Κομισιόν αξιολογεί τις συμβαστικές μας προτάσεις. Μα δεν είναι δικιά μας δουλειά αυτή να σχηματίσουμε άποψη πριν ακούσουμε τις πολύτιμες συμβουλές της Κομισιόν. Ε, είμαι πάρα πολύ ενοχλημένος όσον αφορά αυτή την ε, τοποθέτηση. Καλά αυτό που είπατε, αλλά αφήστε πρώτα να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας ε, καθησυχάζω τους συναδέλφους, ε, οπωσδήποτε θα καταλήξουμε συμβαστικές τροπολογίες, αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα. Ναι, Ισμαήλ Ερτούγαλ, μια ερώτηση. Ε, κοιτάξτε, θα ήθελα να παρακαλέσω τους εκπροσώπους εδώ πέρα της Κομισιόν. Ξέρω πως δεν λαμβάνουν αυτοί τις αποφάσεις, αλλά ε, και εγώ και ο πρόεδρος ε, κάναμε μια ερώτηση και παρακαλώ να διαβιβαστεί. Γιατί δεν δραστηριοποιείται η Κομισιόν. Όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χώρες που δεν εφαρμόζουν ε, την νομοθεσία εν μέρη καθόλου. Και κύριε πρόεδρε καλό είναι και η κυρία Μπούλσο εκεί πέρα να κινηθεί. δεν ξέρω αν έχει και αυτή τη δυνατότητα εν πάση να τα επιβάλλει, αλλά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Γιατί έτσι μόνο θα υπάρχει αποδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρόμπερτ Τσίλε. Ναι, ευχαριστώ. Ο Μάρκους. Και ο Μάρκος ξεκίνησε. Μου έδωσε την πάσα. Από τη διαδικαστική σκοπιά έχει απολύτως λάθος και δεν χρειάζεται να γίνει αυτή η συζήτηση πριν τελευταία συνεδρία των σκιωδών. Οπότε νομίζω πως είναι λίγο λάθος η συζήτηση. Αλλά ευχαριστούμε την Κομισιόν για τις επαγγελματικέ της εξηγήσεις. Γιατί νομίζω πως όλοι μας ε, ενδιαφερόμαστε να έχουμε μια καλή γνωμοδότηση. Αυτά, ευχαριστώ. ευχαριστώ. Κύριε λοιπόν, Κύριο Ντέλη, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν έχω. Σα ευχαριστώ. Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα εδώ πέρα είναι κάποια στιγμή να φύγουμε από αυτόν τον όρο, από αυτή την έκφραση κοινωνικό dumping, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. τα τελευταία χρόνια είχαμε τόσα πολλά αρνητικά για αυτό το όρο τόσο κάποτε πρέπει να τελειώσει αυτή η συζήτηση. Αλλιώς θα συνεχίσουμε να είμαστε διχασμένοι και να αυξάνουν να αυξάνει η αλαζονία. Ευχαριστώ Πέτερ Λούντκριν αλλά σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, είναι κάπως ανησυχητικά αυτά τα οποία ακούμε. Δηλαδή έχουμε την εντύπωση εδώ ότι κανείς δεν ξέρει τι είναι το κοινωνικό ντάμπινγκ. Κοινωνικό ντάμπινγκ σημαίνει να εξαναγκάζουμε τους οδηγούς να οδηγούν με άθλιες συνθήκες να περνάνε ένα μήνα μέσα στο φορτηγό, να τρώνε εκεί, να πλένονται εκεί για να πληρώνται 200 ευρώ το μήνα. Το φορτηγό δεν είναι μέρος για να ζει κανείς. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι δεν ξέρουμε τι είναι κοινωνικό ντάμπινγκ. Τι άλλο περιμένουμε ακόμα δηλαδή. Δεν μπορεί να λέτε ότι δεν ξέρετε τι εστί κοινωνικό τάμπινγκ. Μία ερώτηση μόνο γιατί είπατε ότι δεν ήταν σαφής η νομοθεσία και είναι υπεύθυνα τα κράτη-μέλη. Κοιτάξτε, είναι σαφές για τον χρόνο ξεκούρασης πως πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό ελέγχων των κρατών μελών. Και λέτε πως κάποια κράτη-μέλη είναι στο 0,1% ή δεν ασχολούνται καθόλου με το θέμα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία λοιπόν εδώ πέρα. Εσείς πρέπει να πείτε, είστε υπεύθυνοι, κάνατε κάτι. Τι κάνατε και τι κάνετε για να θυμίσετε ότι και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία πρέπει να τηρείται. Θέλουμε μια ξεκάθαρη απάντηση. Αλλιώς, εντάξει, να ξαναδιορθώσουμε την νομοθεσία, αλλά δεν χρειάζεται, γιατί νομίζω είναι σαφής. Λοιπόν, να σας ακούσουμε και μετά πάλι εισηγηθείς. δύσκολο για μένα να προσθέσω κάτι περισσότερο σε αυτά που είπα προηγουμένως, λέει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Είναι ένα πράγμα για τις ε, αρχές των κάτω μελών να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο ελέγχων και να γίνονται οι έλεγχοι αυτοί, αλλά αν θέλουμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπαίνει στην επικεφαλίδα των διαμεθοριακών συνεργασιών για την εφαρμογή και εδώ αναφέρομαι ιδιαίτερα στο θέμα των εταιριών γραμματοκιβωτίου. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την ανταλλαγή απόψεων και τη δυνατότητα για τα κράτη-μέλη σε ένα κράτος μέρος να ζητούν πληροφορίες από αρχές, σε, από τις ελεγκτικές αρχές άλλων κρατών μελών. Η εφαρμογή δεν είναι μονάχα λοιπόν ένα θέμα ποσοστού των ελέγχων αν θέλουμε να ελέγξουμε τους ελέγχους αυτούς, πρέπει να βελτιώσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό μεταξύ των εφαρμοστικών αρχών. Μερσή λέει ο πρόεδρος και τώρα ο εισήτης, ο κύριος Σνίλσεν που έχει ακούσει όλα αυτά και μπορεί να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Να απαντήσω εφόσον δίναμε. Ήταν μια πολύ καλή συζήτηση και νομίζω ότι ελέγχθηκαν πολλά ευφυή πράγματα. Εγώ είμαι κάπως απεγοητευμένο από την αντίδραση τη Κομισιόν. Εσείς αναφερθήκατε στην δική μας συζήτηση. Καλό είναι αυτό. Φυσικά η Κομισιόν πρέπει πάντα να σχολιάζει τις θέσεις του Κοινοβουλίου. Αλλά μήπως η Κομισιόν θα έπρεπε να απαντήσει καλύτερα τα τεχνικά ερωτήματα τα οποία τέθηκαν αντί να σχολιάζει τις θέσεις του Κοινοβουλίου. Όλοι μας θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα βελτιωθούν οι έλεγχοι Στην Σουηδία έχουμε 2.000 φορτηγά. Σας φαίνεται μικρός ο αριθμός αυτός αλλά ακόμα και στη Σουηδία δεν γίνονται επαρκώς οι έλεγχοι, τότε η Κομισιόν πρέπει να επέμβει και να εξασφαλίσει ότι γίνονται σωστά. Η έλεγχη αυτό είναι η δουλειά της Κομισιόν. Άλλα πράγματα που ελέγχθηκαν. Σας λέω και πάλι, πάλι με απογοητεύει η απάντηση της Κομισιόν και ελπίζω ότι η Επίτροπος Μπούλτς θα μπορέσει να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία έχουμε θέσει. Η πρόταση αυτή λοιπόν τροποποίησης της οδηγίας θα έχει επιπτώσεις στον τομέα αυτό της, ε, των μεταφορών. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτή η οδηγία θα καλύψει τη συγκεκριμένη προβληματική του τομέα του. Τι θα μας προτείνει λοιπόν η Κομισιόν για το τομέα των μεταφορών. Αυτό θέλω να ξέρω. Τι θα κάνει μέσα στην τροποποίηση της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων, ειδικά για το τομέα των μεταφορών. Εδώ θέλουμε να δούμε λοιπόν ποια είναι η... Θέλουμε η Κομισιό να καταλάβει ποια είναι η θέση του Κοινοβουλίου και να τη λάβει υπόψη Και εγώ μπορώ να σας πω μοναχα τι γίνεται στη δική μου χώρα. Δεν είναι θέμα Ανατολής Δύσης. Είναι περισσότερο το θέμα του να μπορούν να μπορεί να συνδυαστεί η εθνική ένωμη τάξη με την εσωτερική αγορά. Γιατί ξέρετε ότι όλες οι χώρες μας έχουν διαφορετικές συνθήκες για τα κοινωνικά θέματα. Είναι διαφορετικές οι κατάσεις, είναι διαφορετικές οι προσεγγίσεις και αυτό πρέπει να εξετάσουμε και θα πρέπει να βρούμε κανόνες ώστε να υπάρχει δυνατότητα του θεμητού ανταγωνισμού σε όλες τις χώρες μας. Δεν θέλουμε αθέμητο ανταγωνισμό, δεν θέλουμε κοινωνικό ντάμπινγκ. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό ο κύριος Γιούγκερ να κατανοήσει επιτέλους ότι θα πρέπει να αναβαθμίσουμε και τον κοινωνικό πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάρουμε στα σοβαρά τα θέματα αυτά. Και η Κομισιόν έχει προετοιμάσει το πακέτο για τα σιδηροδομικά θέματα, όπου πρέπει να ενισχυθεί, πιστεύω, ιδιαίτερα ο κοινωνικός πυλώνας. Πιστεύω λοιπόν ότι και η αυριανή συζήτηση μεταξύ των σκιωδών εισηγητών θα είναι χρήσιμη για να προχωρήσουμε περισσότερο προς την κατεύθυνση μιας κοινή γραμμής ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια σωστή γνωμοδότηση από την πλευρά της Επιτροπής μας, η οποία θα κάνει σαφές ότι λέμε ναι στον θεμητό ανταγωνισμό, αλλά συγχρόνως όχι στο κοινωνικό dumping, ώστε οι αρμόδιες αρχές τα θέματα μεταφορών να μπορούν να παίξουν το ρόλο τους και για τον Ευρωπαϊκό Φορέα που αναφέρθηκε. Όχι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται σε εθνικό επίπεδο οι έλεγχοι, αλλά θα πρέπει η Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι θα γίνονται σωστά σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να έχουν οι εθνικές αρχές την ε, ε, ευθύνη. Ένας ευρωπαϊκός φορέας θα μπορούσε να παίξει ρόλο σε άλλους τομείς ελέγχου. Αλλά πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να πιέσει τα κράτη-μέλη για να είναι πιο αυστηρή ή και καλύτερη η ελέγχη σε εθνικό επίπεδο. Εδώ θα μπορούσε να υπάρχει πράγματι λόγος, για, θα υπάρχει ρόλος για ένα ευρωπαϊκό φορέα ή για τις ευρωπαϊκές αρχές. Προσβλέπω λοιπόν στην αυριανή συζήτηση που θα κάνουμε μεταξύ σκιωδών. Και πάλι. Ευχαριστώ και πάλι τον συγητή για την έκθεση και τη συναρπαστική συζήτηση. Νομίζω άξιζε το χρόνο που αφιερώσαμε ψηφοφορία είναι στις 17 Απριλίου 9 η ώρα το πρωί 5η. Ε, Λίγο τη συνεδρία, τα λέμε στις 3.